Bring the meeting to order. Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Can I do the adoption of the draft agenda first, then I'll come to you, Mike. Εγκρίνεται το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Ο κύριος Κράμερ εδώ πέρα έχει κάτι από τις διαδικασίες. Θα ήθελα αύριο οι συντονιστές να συζητήσουν κάτι γιατί η Κομισιόν θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος ε, του Κοινοβουλίου. Ε, πρόκειται για τα γίγαντο φορτηγά τα οποία απαγορεύονται δια συνοριακά. Και τι γίνεται τώρα, είχα κάνει εγώ μία ερώτηση για μία διαδικασία επί παραβάση. Γιατί δεν επιτρέπεται να πάνε, να περνάνε τα σύνορα. Και αναφέρεται πως έχει απευθύνει ο Επίτροπος ε, μία επιστολή στην Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών πως ερμηνεύει τώρα αλλιώ τον ε, νόμο ε, και λέει θα το επιτρέψει. Καλά, πέρα το ότι εγώ διαφωνώ με τα φορτηγά αυτά, αλλά εδώ πέρα πρόκειται για μια παρανομία της Κομισιόν και θέλω να ζητήσω από τον Επίτροπο να μην ε, γράψει, ε, να μην ε, στείλει αυτή την επιστολή και θα ήθελα να παρακαλέσω και σένα, Μπραν Σίμψον, να το υπενθυμίσεις στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου που είπε πως πρέπει το Κοινοβούλιο επιτέλους να το παίρνει σοβαρά ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου θέματος πως δεν θα πρέπει να αποσταλεί αυτή η επιστολή δεν είναι δυνατόν να παραβιάζει την ε, νομοθεσία ο Επίτροπος ε, αδιαφορώντας τελείως για το Κοινοβούλιο Σας ευχαριστώ όπως ξέρετε μίλησα με τον Επίτροπο και ανέφερα το θέμα τη θέση της Επιτροπής μας μου έδωσε την εξήγηση που μου δώσατε κι εσείς για το ότι νομικά λένε πως είναι εντάξει το έχω βάλει στην ημερήσια διάταξη για τη συνεδρία των συντονιστών στα διάφορα θα το συζητήσουν λοιπόν αύριο οι συντονιστές προτείνω να το συζητήσουμε τότε και βεβαίως αυτή η απόφαση ε, ούτως ή άλλως θα πρέπει να επικυρωθεί από την Επιτροπή στο σύνολό της Τετάρτη. Ναι, κύριε Κράμερ, κάτι ακόμα. Ε, να σας αναφέρω τι μου είπαν ακριβώς. Για ε, προσπάθειες διάσκησης των συνόρων από τέτοια φορτηγά δεν ενημερώθηκε η Κομισιόν. Εάν η Κομισιόν ενημερωνόταν για κάτι τέτοιο θα ε, ζητούσε διευκρινήσεις από το εν λόγω κράτος μέλος ή κράτης μέλης. Εάν δεν ε, επενέβαιναν για την απαγόρευση αυτών των ορμολογίων τα κράτη μόλι, η Κομισιόν θα κινούσε διαδικασία ε, επί παραβάση. Αυτή ήταν απάντηση που μου έδωσαν ε, αρχές ε, Φεβρουαρίου, νομίζω 2012. Ναι, ναι, μα το είδα και εγώ. Προτείνω να το συζητήσουμε οι συντονιστές αύριο και μετά ότι και να αποφασίσουμε θα το υποβάλουμε στο σύνολο της Επιτροπής. Δεν έχω δικαίωμα να απευθύνω βεβαίως επιστολή πριν ε, με εξουσιοδοτήσει η Επιτροπή. Αλλά αυτό το οποίο είπατε νομίζω πως το ακούει η Κομισιόν, οπότε οπωσδήποτε θα φτάσει στα αυτιά του Επιτρόπου. Οπότε και εγώ ε, θα συναντηθώ απόψε με την Κομισιόν για να τους μεταφέρω αυτά που τους είπα και το Σώτο Κυριακό. Ωραία. Περνάμε λοιπόν στην έγκριση των πρακτικών της συνάντησης της 6 Φεβρουαρίου. Συμφωνείτε όλοι? Α, ναι μπορώ να περάσω στο μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και αερομεταφορών, έκθεση Bradburn, εξέταση τροπολογιών. Να υπενθυμίσω, Φίλιπ, στους ε, βουλευτές πως η ευριανή ψηφοφορία αναβλήθηκε για τον Μάρτιο. Οπότε θα εξετάσουμε απλά τις τροπολογίες. Δεν θα έχουμε ψηφοφορία αύριο. Σωστά, κύριε Μπράντον. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως στην επόμενη συνεδρία θα γίνει ψηφοφορία. Και αυτό γιατί είναι πολλές οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και, έχουμε και την, είχαμε και την πράσινη εβδομάδα. Επομένως, θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να λάβουν τις τροπολογίες μετεφρασμένες και να μπορέσουν να τις διαβάσουν, να τις μελετήσουν. Θα ήθελα να κάνω ένα-δύο σχόλια για τις τροπολογίες, ε, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα εξετάσω την κάθε μία ξεχωριστά. Θα ήθελα απλώ να σας πω ότι εν γέννη είναι πολύ χρήσιμες οι τροπολογίες αυτές. Υπάρχουν κάποιες ε, συγκεκριμένες τροπολογίες ε, για τις οποίες έχω κάποιες αμφιβολίες γιατί δεν έχουν να κάνουν με τα περιφερειακά αεροδρόμια. Είναι λίγο πιο γενικές ε, οι τροπολογίες αυτές. Επομένως βγαίνουν κάπως από το πεδίο εφαρμογή ε, τη ε, έκθεση αυτή. Πάντω οι τροπολογίε είναι πολύ χρήσιμε. Θα συναντηθώ με του σκιώδει ηγητέ την ε, Τετάρτη και θα προσπαθήσω να καταλήξω σε κάποιε συμβαστικέ τροπολογίε. Του των ευθέτων, κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήθελα να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, να αναφερθώ σε, κάποια βασι... σε κάποιες βασικές θεματικές κατηγορίες των τροπολογιών αυτών. Αν δούμε καταρχάς τα εκτιμώντας. Εκεί πέρα είχαμε ορισμένε ε, τροπολογίες από τον κύριο Ούτζας, ε, από τον κύριο Σασόλη επίσης. Έχουμε κάποιες χρήσιμες λοιπόν τροπολογίες όπου προσπαθούμε να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο περιφερειακό αεροδρόμιο, περιφερειακό αερολιμένα. Στην αρχική μα συζήτηση το είχαμε πει, κύριε Πρόεδρο, ότι είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να ορίσουμε τα αεροδρόμια αυτά και τι σχετικέ υπηρεσίε. Πολύ συχνά αναφερόμαστε απλώ σε κάποια αριθμητικά δεδομένα και αυτό δεν μα βοηθά να συνειδητοποιήσουμε τι είναι τελικά ένα περιφερειακό αεροδρόμιο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να έχουμε μια πιο ένα, καλύτερο ορισμό, μια καλύτερη αιτιολογία και οι τροπολογίε οι σχετικές που λάβαμε θα μα βοηθήσουν να καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική τροπολογία. Δεύτερη κατηγορία όσον αφορά τι υποχρώσεις των δημοσίων υπηρεσιών και τι κρατικέ βοήθειε και ενισχύσει. Πάλι εδώ πέρα είχαμε χρήσιμε τροπολογίε από διάφορου συναδέλφου για το ζήτημα αυτό και πάλι ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική τροπολογία όσον αφορά το ζήτημα του One Bag Rule. Θα θέλω προς αυτό να πω κύριε Πρόεδρε ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα με κάποιες ε, αεροπορικές εταιρείες ε, low cost όπου ε, έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τις αεροπορικές αυτές εταιρείε. Πρέπει όμως να ασχοληθούμε πιο συγκεκριμένα με τα περιφερειακά αεροδρόμια και με τις περιφερειακές αεροπορικές υπηρεσίες. Να μην υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα όρια όσον αφορά τις αποσκευές που μπορεί να έχει μαζί το επιβάτης, ιδίως όταν χρησιμοποιείται ένα μικρό περιφερειακό αεροδρόμιο, γιατί αναγκαστικά εκεί θα χρησιμοποιηθεί και ένα μικρό αεροσκάφος. Και ξέρετε ότι πολύ συχνά οι επιβάτες έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί φτάνουν στο αεροδρόμιο, έχουν μία αποσκευή και ξαφνικά τους λένε στο αεροδρόμιο πια ότι η αποσκευή αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή, γιατί είναι πολύ μικρότερο σκάφος. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένους ορισμούς για το τι είδους αποσκευές μπορούν να έχουν οι επιβάτες σε ένα μικρό αεροσκάφος, το οποίο έχει μικρότερη βέβαια χωρητικότητα. Έχουμε λοιπόν κάποιες σχετικές τροπολογίες και πιστεύω ότι και με αυτές θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική τροπολογία. Το επόμενο ζήτημα όπου είχαμε πάλι αρκετές τροπολογίες, κυρίως από τον κύριο Πέρκερ, τον κύριο Ουτζέσσα και άλλους συναδέλφους, έχει να κάνει με τις διατροπικέ συνδέσει και αυτές οι τροπολογίες είναι πολύ χρήσιμες. Θέλουμε ουσιαστικά στην έκθεση αυτή να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πολυτροπικές ε, διασυνδέσεις ανάμεσα στα περιφερειακά αεροδρόμια και άλλα μέσα και άλλους τρόπους μεταφοράς και οι τροπολογίες αυτές μας βοηθούν να το πετύχουμε αυτό. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να αφαιρθούμε στη γενικότερη επίπτωση των περιφερειακών αεροδρομίων για τις οικονομίες ε, σε επίπεδο περιφέρειας. Υπάρχουν πάλι και εδώ πέρα κάποιες τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στη συμπερίληψη κάποιων μεγαλύτερων περιφερειακών αεροδρομίων στο κεντρικό δίκτυο διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Υποστηρίζω τις α, τροπολογίες αυτές και πραγματικά μπορούν να δώσουν μια καλύτερη όθηση οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και μια, μια καλύτερη ενθάρρυνση για την ανάπτυξη περιφερειακών αερολιμένων και αεροπορικών σχετικών υπηρεσιών. Έλαβα, όπως σας είπα, πολλές τροπολογίες θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για τις ε, τροπολογίες αυτές, οι οποίες ως επιτοπλίστων ιδιαίτερα χρήσιμε. και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε την Τετάρτη να καταλήξουμε σε κάποιες καλές συμβαστικές τροπολογίες, προκειμένου να ψηφίσουμε στην επόμενη μα πλέον συνεδρίαση την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. E, Ο Πέρκερ, εξ του ΕΛΚ. Äh, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είχαμε ήδη τη δυνατότητα να συζητήσουμε γενικά την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ τον κύριο Μπράντμπεν για την ε, συνεργασία που είχαμε πριν ε, ακόμα τη σύνταξη της έκθεσης και συνεχίστηκε μέχρι την ε, προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια γραμμή ψηφοφορίας για τις πολλές ε, τροπολογίες. Θα υποστηρίξω εγώ τον ε, κύριο Μπράντμπερν ε, στο κομμάτι αναζήτησης μιας διεξόδου για τις κρατικές ενισχύσεις γιατί εδώ πέρα πρέπει να το συζητήσουμε για το εάν πράγματι ο δημόσιος τομέας πρέπει ή επιτρέπεται να στηρίζει έτσι τα περιφερειακά αεροδρόμια για να διατηρήσουν την κυκλοφορία εκεί πέρα. Εδώ σας παραπέμπω σε έναν έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια έρευνα που αφορούσε αεροδρόμια στη Γερμανία και στην ε, Αυστρία που συμπεριλάμβανε και το αεροδρόμιο του Κλάγκενφουρτ του τόπου μου όπου ασκήθηκε σοβαρή κριτική στο ότι έχουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μέσω του ότι ο δημόσιος τομέας οδηγεί σε κάλυψη του κόστους που έχουν οι αεροπορικές εταιρείες. Και είναι απαράδεκτες αυτές οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Και μιλάμε ακριβώς για τα αεροδρόμια που θα υπάγονται στον, στο θέμα μας εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να βρούμε κάποιους άλλους τρόπους για να γίνουν ξανά πιο ελκυστικά αυτά τα αεροδρόμια από όσο είναι αυτή τη στιγμή. Προβληματικό θεωρώ και θέλω να το πω την περιορισμένη κατά την άποψή μου σκοπιά που έχουμε εδώ πέρα. Όταν μιλάμε για τα προβλήματα των περιφερειακών αεροδρομίων, για τον κανονισμό της μίας αποσκευής. Ε, ε, αυτό που εισήχθη είχε οδηγήσει σε 65% μείωση των ε, επενδύσεων. Ε, μου φαίνεται λοιπόν πως ε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες μάλλον που προκάλεσαν αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω αν φταίει μόνο ένας κανονισμός. Για τα αεροδρόμια αυτά, τα οποία όπως είπαμε είναι πολύ σημαντικά για πολλές περιφέρειες. Οι ε, τροπολογίες του ΕΛΚ αναφέρονται λίγο ή σε μέτρα τα οποία πάνε στην τάση ότι όλα θα τα πληρώνει ο φορολογούμενος. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε μία συμβιβαστική ε, λύση. Ε, αυτό είναι κάτι παρόμοιο με το κόστος ε, του ελέγχου ασφαλείας όπου είναι δυσανάλογο και πάλι το επομίζεται ο φορολογούμενος. Δεν γίνεται κάθε φορά όλα αυτά τα προβλήματα να τα πληρώνει ο φορολογούμενος. Πρέπει να βρεθούμε άλλους, ε, πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Ε, ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα μικρά αεροδρόμια ως αεροδρόμια με τα οποία θα αποφεύγει κανείς τα μεγάλα στα οποία δημιουργείται πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Αλλά δεν ξέρω βέβαια θα πρέπει να δούμε και σε τι αποτελέσματα οδηγεί αυτό. Ε, θετικό είναι επίσης το ότι τονίζεται ο συνδυασμός μέσων μεταφοράς και πράγματι ασκείται σωστή κριτική στο ότι υπάρχουν καθυστερεί στο ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Αυτό βεβαίω είναι ένα γενικό πρόβλημα, δεν αφορά μόνο τα περιφερειακά αεροδρόμια. Συνοψίζοντας λοιπόν, ελπίζω να ενσωματωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες τροπολογίες σε συμβαστικές τροπολογίες ε, ειδικά δε όσον αφορά το τι πρέπει να κάνει το κράτος να βρούμε μια κοινή προσέγγιση και να μην πληρώνει μόνο φορολογούμενος για να στηρίξουμε και σημαντικά περιφερειακά αεροδρόμια για να μπορούν να επιτελούν τη λειτουργία τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Σασόλη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπράντμπορν για την ε, εργασία του και επειδή έλαβε υπόψη τις ε, προτάσεις που προέβαλα ως κοιόδης εξ των σοσιαλιστών. Θα ήθελα να εκφράσω δύο σκέψεις σε ορισμένα σημεία που κατά τη γνώμη μου μπορούν να βελτιωθούν. Το πρώτο αφορά την τροπολογία συμβιβασμού 1. Γνωρίζω ότι όταν μιλάμε για ορισμό περιφερειακού αεροδρομίου, ο ορισμός αυτός είναι δύσκολος. Στο συμβιβασμό προτείνεται εκ νέου ο ορισμός ενός ε, αεροδρομίου που είναι non-hub, που δεν είναι κομβικό δηλαδή. Και αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι να λάβουμε υπόψη μερικές μεταβλητές οι οποίες αποκλείονται από το συμβασμό όπως η τυπολογία σύνδεσης, τις συνδέσεις με τις πόλεις και τα βασικά αεροδρόμια, καθώς και τον όγκο μεταφοράς τον αριθμό επιβατών δηλαδή. Γι' αυτό θα ήθελα να λάβετε υπόψη την τροπολογία υπαριθμών 1 που ελήφθη υπόψη για το συμβιβασμό υπαριθμών 1. Δεύτερον, σας ευχαριστώ πολύ διότι λάβατε υπόψη την τροπολογία 39 στο Συμβασμό 5, δηλαδή τις κρατικές επιδοτήσεις ως προς τους περιφερειακούς αερολιμένες που είναι ζωτική σημασία για πολλές περιφέρειες. Πιστεύω ότι ο κρατικός μηχανισμός και η διοίκηση υποστηρίζουν άμεσα ή έμεσα μία εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη την περιφέρεια, την ελόγω περιφέρεια. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τις άμεσες ή έμεσες επιδοτήσεις, αλλά δεν ξέρουμε πόσο ισχύει αυτή η δέσμευση. Γι' αυτό κατά την άποψή μου θα πρέπει να συνδέσουμε περισσότερο τη δέσμευση των ε, αερομεταφορών, των, ε, δηλαδή των αεροπορικών γραμμών σε σχέση με τη διάρκεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, η δημόσια η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να επαληθεύσει και να προβεί σε έρευνες ως προς το αεροδρόμιο, το περιφερειακό, το περιφερειακό αερολιμένα, αυτό μπορεί να έχει και μειονεκτήματα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, γι' αυτό θα ήθελα στην τροπολογία συμβασμού 5 να εντάξετε τη δική μου 39 που ζητά σχέση αναλογικότητας μεταξύ των κρατικών επιδοτήσεων και του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μία εταιρεία πρέπει να παραμείνει στο αεροδρόμιο υποχρηματοδότηση. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον, ε, και τον αριθμό των επιβατών, τον όγκο διέλευσης όπως ορίζεται. Τέλος, θα ήθελα να πω προς τους Ιταλούς συναδέλφους ότι στην 77 υπάρχει ένα λάθος στη μετάφραση. Όπως είδαμε με τους υπαλλήλους της Επιτροπής, δεν έχει ενταχθεί το πρώτο μέρος της τροπολογίας μου και γι' αυτό θα ήθελα να σας αποστείλω το πλήρες κείμενο. Ευχαριστούμε κύριε Σασόλη και κυρία Μάισλε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μιλώ εξ ονόματος του κυρίου Ούτζας. Ζητά συγγνώμη γιατί δεν μπορεί να παρευρεθεί για απρόβλεπτους λόγους και θα ήθελα να ευχαριστήσει τον κύριο Μπράντμπουρν για την εξαιρετική εργασία και για τις προτάσεις συμβιβασμού που ήταν ένα καλό σημείο εκκίνησης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ευχαριστεί και τον εισηγητή, διότι έλαβε υπόψη αρκετές υποδείξει ως προς τους συμβασμούς 4 και 9. Έχει και ορισμένε παρατηρήσεις και τώρα θα σας διαβάσω τι μου έγραψε. Ως προς την ε, πρόταση συμβιβασμού 1, σε σχέση με τον ορισμό των ε, περιφερειακών αερολιμένων που συζητήθηκε, θεωρώ ότι η τροπολογία δεν είναι ικανοποιητική. Γνωρίζω ότι πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα και θα ήταν δύσκολο να φτάσουμε σε μια συμφωνία μεταξύ όλων των συμβαλωμένων μερών, τότε θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια για να αναγνωρίσουμε ορισμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά που είναι κοινά για τους περιφερειακούς αερολιμένους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υφίσταται ο ορισμός ή να μιλήσουμε για μη κομβικούς αερολιμένες. Γι' αυτό όρισα ένα προσχέδιο πρότασης τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ ε, μεγάλων μιζώνων και ε, ελασσόνων αεροδρομίων και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει τα, τους περιφερειακούς αερολιμένες λαμβάνοντας υπόψη τι ε, σχέσεις συνδεσιμότητας υπάρχουν, δηλαδή κυρίως όγκος διέλευσης. Ελπίζω όλοι οι συνάδελφοι να λάβουν υπόψη αυτές τις υποδείξεις. Ως προς το, την πρόταση Συμβασμού 8, ίσως αναφέρεται στις χρονοθυρίδες που ζητήθηκαν από έναν Βρετανικό φορέα το καλοκαίρι του 2011. Διενεργήθηκε μία μελέτη λοιπόν και θεώρησε ότι οι περιφερικοί αερολιμένες δεν πλήττονται από τη συμφόρηση ή χαμηλή χωρητικότητα. Δεν χρειάζονται καν έναν συντονιστή για την κατανομή χρονοθυρίδων. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εντελώς λανθασμένη η αναφορά σε αυτή τη μελέτη και θεωρώ ότι θα πρέπει να διαγραφεί η μνήμα που αφορά την κατανομή χρονοθυρίδων. Επίσης έχω υποβάλει και άλλες τροπολογίες πέρα από τους συμβιβασμούς και θα ήθελα να υποστηρίξετε στις 47 και 52. Η 47 τονίζει τη συνδεσιμότητα μεταξύ περιφερειακών αερολιμένων και τουριστικού τομέα που αφορά την Ιταλία και ζητούμε ώστε οι συμβατικοί αυτοί όροι να ισχύσουν ιδιαίτερα όπου υπάρχουν εταιρείε χαμηλού κόστου. Στη 52 γίνεται λόγος για διαχείριση περιφερειακών αερολιμένων με την κατάλληλη υποδομή και με τις ε, ε, διαφοροποιήσεις και αλλαγές έτσι ώστε όλοι οι επιβάτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα σημεία του αερολιμένα. Αυτά μου ζήτησε να σας διαβάσω ο κύριος Σούτζας. Ε, ως προς τα, το κατατάλα, την κατά πολύ καλή έκθεση, ο κύριος Κράμερ. Ναι. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ καθυστέρησε με το αεροπλάνο αλλά αυτό είναι καθημερινό γεγονός πια. Κάποιος συνέχεια ε, πρέπει να απουσιάζει. Δεν ξέρω τώρα κάποια τεχνικά προβλήματα. Βεβαίω θα ήθελε και εκείνη να ευχαριστήσει τον εισηγητή, αν και δεν συμφωνεί με όλα, γιατί όπως ανέφερε και ο συνάδελφος πριν, για, τα, για τη δημόσια χρηματοδότηση για τα αεροδρομία να πω πως κάθε χρόνο ο Ευρωπαίος φορολογούμενος πληρώνει 30 δισεκατομμύρια σε αεροπορικές εταιρείε γιατί δεν υπάρχει φόρο στα καύσιμα των αεροσκαφών. 30 δισεκατομμύρια ευρώ αν πήγαιναν στους σιδηροδρόμους θα είχαμε φοβερά δίκτυα με χαμηλές ε, τιμές. Οπότε δίνουμε σε λάθος μέρος τα δημόσια κονδύλια. Βεβαίως, στα περιφερειακά αεροδρόμια υπάρχουν κάποια αεροδρόμια που πρέπει να διατηρηθούν, ακόμα και αν δεν ε, αποδίδουν οικονομικά, π.χ. σε νησιά. Εκεί πέρα είναι υποχρεωμένο το κράτος να τα στηρίξει. Αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Π.χ. στη Γερμανία δεν είναι η αρμοδιότητα για την αεροπορία ομοσπονδιακή, αλλά σε κάθε κρατήδιο. Και τα κρατήδια τσακώνονται το ένα με το άλλο. Π.χ. τα αεροδρόμια του Ζαρμπρίκεν και του Βαϊμπρίκεν. Μιλάμε για αεροδρόμια που απέχουν 60 χιλιόμετρα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, η μόνη σύνδεση που υπάρχει είναι τρένο, δεν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά το κάθε κρατήδιο θεωρεί πως πρέπει να έχει δικό του αεροδρόμιο. Και γίνονται και κόλπα. Λέει η πόλη του Ζαρμπρούγκεν πως θα έχουμε 900 πτήσεις το χρόνο, αλλά βεβαίως 900 ε, ε, από αυτές τις φορές ε, δεν γίνονται οι πτήσεις. Όλα αυτά με κόστος του φορολογούμενου. Κάναμε λοιπόν, υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες, κάποιες έγιναν δεκτές, κάποιες ε, άλλες όχι. Χρειαζόμαστε λοιπόν δίκαιο ανταγωνισμό, όχι μόνο στα κάψιμα, αλλά και... Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για δημόσιες ενισχύσει. είτε θα ισχύει για όλα τα μέσα μεταφοράς ή για κανένα. Δεν μπορεί ε, να κλείνουν σιδηρόδρομοι γιατί δεν αποδίδουν, αλλά να προωθούμε τις αεροπορικές εταιρείε. Δεν είναι δυνατόν. Επίσης δεν είναι δυνατόν να έχουμε διαφορετικό σύστημα τιμολόγησης. Γιατί ξέρετε η Γερμανία έχει 19% φόρο στις διεθνείς ε, πτήσεις ε, και λίγα κράτη-μέλη έχουν τόσο υψηλό φόρο, αλλά υπάρχει και το πρόβλημα της μετάβασης από το σιδηρόδρομο στο αεροπλάνο και πρέπει να δούμε τη σύνδεση με τους σιδηροδρόμους. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε το λάθος, το ότι στη Γαλλία έχουμε 10 νέους ε, σταθμούς ΤΖΒ ε, που δεν συνδέονται με τα αεροδρόμια και χάνει το χρόνο που έχει κερδίσει κανείς με το τρένο. Εάν ε, αποδίδουν τα, αεροδρόμια θα πρέπει να συνδεθούν οπωσδήποτε. Και βεβαίως ο έλεγχος των υγρών στα αεροδρόμια καταστροφή, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, μόνο καψώνει. Είναι, για, παριστάνουν ότι κάνουν κάτι και δεν μπορεί κανείς να διαπιστώσει βεβαίως αν είναι επικίνδυνο το υγρό ή όχι. Ε, αν είναι, αν χρειάζομαι όντως ε, κάτι, κάποιο υγρό για να κάνω το εκρηκτικό, πάω και το αγοράζω μετά, αφού περάσω από τον έλεγχο από τα duty free. Ε, δεν έχει κανένα νόημα λοιπόν αυτός ο κανονισμός. Οπότε θα είναι δίκαιο ανταγωνισμό για όλα τα μέσα μεταφορά. Ευχαριστώ. Αν θέλετε να μιλήσετε για αυτό το θέμα, σας παρακαλώ ε, να μας ειδοποιείτε, κύριε Κόλτσακ, για να, για να το βλέπουμε. Εάν το ζητήσετε από την αρχή, βοηθάει και εμένα να είμαι και δίκαιος με την κατανομή του χρόνου. Όταν έρχονται αργά οι συνάδελφοι, ε, μειώνει το χρόνο που έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε θα σας παρακαλούσα πολύ ε, να ζητά το λόγο εξ να βοηθήσετε και το, τον πρόεδρο. Θα ήθελα να πω ότι ο εισηγητής έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους μου. Και που και που, αυτή τη φορά τουλάχιστον, συμφωνώ με τον συνάδελφο από τους Πρασίνους. Προτιμάμε να έχουμε αυτή τη μορφή μεταφορών σε σχέση με άλλες, ιδίως όσον αφορά τα περιφερειακά αεροδρόμια, έχει απόλυτο δίκιο. Κύριε Μπράτμπορν, σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Σας ευχαριστώ επίσης για τι συμβαστικέ τροπολογίες, τι οποίε καταλήξατε, στι συμφωνίες με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Μπράντβερν. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, αυτή η απέτηση από τα κράτη-μέλη για τη διασύνδεση των διαφορετικών μέσων μεταφοράς είναι σημαντική αυτή και για τη συμβαστική λύση 7 θεωρώ πως η ποιότητα των υπηρεσιών και των συνθήκων εργασίας είναι κάτι που πρέπει να ξαναδούμε γιατί αυτό δεν σχετίζεται οπωσδήποτε με τον κανονισμό της μίας αποσκευής, αλλά γενικά ε, με τις συνθήκες εργασίας στα αεροδρόμια. Και θεωρώ πως ε, θα πρέπει να έχουμε, νομίζω, ευκαιρίες να το ξανασυζητήσουμε με τον εισηγητή. Επίσης, όσον αφορά το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του βασικού δικτύου και του δευτερεύοντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αλχα Χαντραβή. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θα τονίσω δύο πράγματα που ανέφερε και ο κύριος ε, Σασόρη. Πρώτα απ' όλα, Σασόλη. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό πράγματι να υπάρχει διασύνδεση με ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ όλων των αεροδρομίων και σε κάποια περιφερειακά αεροδρόμια βλέπουμε την παρουσία μιας μεγάλης εταιρείας η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στις τοπικές αρχές και στα αεροδρόμια και έχει πάρα πολλά προνόμια, στήριξη, αλλά μπορεί να απειλήσει και να φύγει από εκεί και έχει έτσι με αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στη λειτουργία του αεροδρομίου. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε για τέτοιες περιπτώσεις και να το αναφέρουμε στην έκθεση. Σε σχέση με αυτό, να συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπαχ, ότι δηλαδή πρέπει να δούμε και τις κοινωνικές πτυχές, τους κανόνες του παιχνιδιού που πρέπει να τηρούνται και στα περιφερειακά αεροδρόμια και από τις εταιρείε χαμηλού κόστους όταν μιλάμε για ίσους όρους ανταγωνισμού. Το δεύτερον ε, που θέλω να τονίσω είναι πως υπάρχει πράγματι μια σχέση με την άλλη έκθεση για τα δικαιώματα των επιβατών, γιατί χρησιμοποιούν αυτά τα αεροδρόμια οι εταιρείε χαμηλού κόστους και ασκείται έτσι κριτική στο πώς ε, συμπεριφέρονται στους επιβάτες. Και πρέπει έτσι να αναφέρουμε κάποια πράγματα. Έχουμε το ζήτημα των ε, αποσκευών και των περιορισμών Οπότε θα πρέπει να έχουμε πιο υποχρεωτικούς κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεύτερο και τελευταίο διαφάνεια στις τιμές. Ξέρετε πως οι εταιρείε χαμηλού κόστους έχουν μετά διαφόρων ειδών ε, χρεώσεις. Φαίνεται μια αρχική χαμηλή τιμή και μετά προστίθενται διάφορα πράγματα. Οπότε πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό. Συνοψίζοντας λοιπόν, στηρίζουμε την έκθεση, αλλά ελπίζουμε να μπορέσουμε να στηρίξουμε και κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω πολλά από τα επιχειρήματα που ακούσαμε από τους συναδέλφους. Θα ήθελα να πω ότι με τις τροπολογίες αυτές προσπαθήσαμε πρώτον να μιλήσουμε για την ολοκλήρωση των δικτύων περιφερειακών αεροδρομίων και θεωρώ ότι η κρίση δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μία χαρτογράφηση των ε, περιφερειακών αερολιμένων έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να μην υπάρχει συμφόρηση ή όταν υπάρχει να την αντιμετωπίσουμε και να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά στο δίκτυο TEN-T. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αρχές εξειδίκευσης, ποιότητας υποδομών και διατροπικότητας Επίσης ε, δίνουμε μεγάλο βάρος και στις μεταφορές ε, φορτίων και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν βελτιώσεις και στους θερματικούς σταθμούς. Επίσης οι κακές πρακτικές όπως η μία χείρα αποσκευή να αντιμετωπιστούν διότι αυτό είναι ασύμβατο με τις προσπάθειες που καταβάλουν πολλά περιφερειακά αεροδρόμια να ανταποκριθούν. Υποβάλλω ορισμένες τροπολογίες συμβιβασμού έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις μειονεκτούσες περιοχές και τέλος Επειδή ακριβώς ο συνάδελφος ε, Τρεμόσα δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ σήμερα για λόγους συμφόρης σε ένα αεροδρόμιο, ότι θα πρέπει να έχουμε σωστή διαχείριση των περιφερειακών αερολιμένων. Θα πρέπει να γνωρίζουμε την ε, τοπική πραγματικότητα που ξέρουν αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά Πιστεύουμε ότι έτσι θα είναι ε, βιώσιμη υποστήριξη των περιφερειακών αεροδρομίων και το πρότυπο αυτό επιτυχίας που υπάρχει να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Διότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες όπου τα περιφερειακά αεροδρόμια την χάνουν διαχείριση από ένα κεντρικό φορέα. Και αυτό δεν είναι το καλύτερο ή το πιο αποδοτικό. Βλέπουμε ότι αυτός ο συγκεντρωτισμός διαχείρισης δεν είναι αποτελεσματικός και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις απομακρυσμένες περιφέρειες. Επίσης υποστηρίζω τις τροπολογίες της Ινέσα Γιάλα και του κυρίου Ούτζας θεωρώ θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση για άτομα με χαμηλότερη, περιορισμένη κινητικότητα. Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπράτμπορν, γιατί η έκθεση του είναι ιδιαίτερα πλήρης. Και νομίζω ότι η αρχική έκθεση, ήδη πριν τις τροπολογίες, κάλυπτε όλα τα βασικά σημεία και νομίζω ότι έρχεται την κατάλληλη στιγμή η έκθεση αυτή. Όχι μόνο επειδή έχουμε το αεροδρομικό πακέτο και άλλα σχετικά νομοθετήματα. Για λόγους διευκρίνησης τώρα, υπάρχουν δύο ξεχωριστά ζητήματα για μένα όσον αφορά το ζήτημα της μία χειραποσκευής. Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να δείξουμε έχει να κάνει με τα αεροδρόμια. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα κάποια αεροδρόμια τα οποία επιτρέπουν ε, επιβάτες με μία μόνο αποσκευή να περάσουν από τα συστήματα ασφαλείας, από τον έλεγχο. Θυμάστε όταν είχαμε τρομοκρατικές απειλές πριν από μερικά χρόνια, όλα τα αεροδρόμια ακολούθησαν τον κανόνα αυτό. Και αυτό προκαλεί αυτή τη στιγμή σύγχυση είναι ότι στη συνέχεια υπέρχαν πολλά αεροδρόμια τα οποία επανήλθαν στον αρχικό κανόνα, δηλαδή των δύο χειραποσκευών, όπου η δεύτερη μπορεί να είναι ένα υπολογιστή ή κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν εμφανίζονται οι επιβάτε με τι ε, χειραποσκευέ του, δεν μπορούν να περάσουν τελικά τη χειραποσκευή μαζί με μια άλλη αποσκευή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, τι γίνεται στη συνέχεια με την αεροπορική εταιρεία και όταν αυτή λαμβάνει μια σχετική απόφαση. Πιστεύω ότι οι αεροπορικέ εταιρείε μέσω των ιστοσελίδων του θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση, τι επιτρέπεται δηλαδή και τι δεν επιτρέπεται στα αεροσκάφη του. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε τουλάχιστον του επιβάτε όταν λαμβάνουν μια απόφαση για το τι θα πάρουν μαζί του. Συμφωνώ επίση με του συναδέλφου στο ακόλουθο σημείο οι περισσότεροι από τον κλάδο δεν συνειδητοποίησαμε ποτέ ότι μία τσάντα με αδοσμολόγητα προϊόντα, με duty free, αποτελεί μία επιπλέον χειραποσκευή. Πολύ συχνά πρόκειται απλώς για μία πλαστική σακούλα που έχει απλώς κάποια αντικείμενα μέσα. Ουδέποτε εγώ θεώρησα ότι αυτή η σακούλα θα μπορούσε να αποτελέσει χειραποσκευή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και το ζήτημα αυτό και πρέπει να εξετιστεί και από αυτού οι οποίοι πρέπει να λάβουν τη σχετική απόφαση για το αν τελικά είναι χειραποσκευή ή όχι. Όσον αφορά τώρα τα PSOs. Σαφώς είναι πολύ σημαντικά σε ορισμένε περιπτώσει δεν θα έχουμε συνθήκε ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, μπορούμε να φανταστούμε ένα περιφερειακό αεροδρόμιο σε ένα νησί όπου μία μόνο αεροπορική εταιρεία εκτελεί πτήσει εκεί. Νομίζω ότι και εκεί πέρα δεν τίθεται ζήτημα κρατικών ενισχύσεων. Το ζήτημα αυτό έχει επιληθεί άλλωστε και στο παρελθόν. Τέλο, όσον αφορά τον ορισμό του περιφερειακού αεροδρομίου. Τι είναι τελικά περιφερειακό αερολιμένας. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αναλώσουμε πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Ο ορισμό ενό περιφερειακού αερολιμένου είναι ο αερολιμένα που βρίσκεται βασικά σε μια περιφέρεια και ένα αεροδρόμιο το οποίο προφανώ είναι μικρότερο από το αεροδρόμιο τη Φραγκφούρτη ή από το Σαλτεγκόλ αλλά σε ορισμένε περιπτώσει μπορεί να έχουμε περιφερειακό αεροδρόμιο, το οποίο να είναι παράλληλα και διεθνέ αεροδρόμιο, όπω για παράδειγμα στο Μάντζεστερ. Ενδεχομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πρέπει να ασχοληθεί λίγο με το ζήτημα αυτό. Και μια τελευταία παρατήρηση για το πόσε αποσκευέ μπορεί να πάρει κανεί μαζί του μέσα στο αεροσκάφο. Μα ξέρετε ότι δεν πρόκειται καν για μια απόφαση η οποία είναι καθαρά εμπορική. Εξαρτάται και από το ίδιο το αεροσκάφος τελικά. Αν υπάρχει απαραίτητη χωρητικότητα μέσα στο αεροσκάφος προκειμένου να πάρει τις αποσκευές αυτές. Τεχνικό λοιπόν το ζήτημα αυτό. Και μια τελευταία παρατήρηση τώρα. Ναι κύριε Μπράντμπορν, η έκθεσή σας θεωρώ ότι είναι πολύ καλή και νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μιλάμε απλώ για τα περιφερειακά αεροδρόμια, μιλάμε για όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, μιλάμε για τον κλάδο του τουρισμού, μιλάμε για τον κλάδο τη αεροναυτιλία και όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε πολύ καλά ζωτικά περιφερειακά αεροδρόμια. Πρέπει και αυτά βέβαια να γίνουν πιο ελκυστικά και ενδεχομένως θα πρέπει να ασχοληθούν λίγο περισσότερο για το λόγο αυτό με το ζήτημα της κοστολόγησης και το ζήτημα των τελών. Προφανώς πρέπει να επιβιώσουν τα αεροδρόμια αυτά, πρέπει να ενθαρρύνουμε τα περιφερειακά αεροδρόμια και θεωρώ ότι ο κύριο Μπράντμπρον έχει καταλήξει σε κάποιε πολύ καλέ συμβαστικέ τροπολογίε, αλλά ούτω ή άλλω από την αρχή η απο ήταν εξαιρετική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριο Χίγκιν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω ξανακούσει άλλη εκθέση να την χάνει τόσο ευρεία αποδοχή. Νομίζω πω είναι εξαιρετική έκθεση. Εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια με τέσσερα περιφερειακά αεροδρόμια που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομία μα, ειδικά όσον αφορά τον τουρισμό στον οποίο βασιζόμαστε. Και νομίζω πω είναι ουσιαστική σημασία να στείλει ένα μήνυμα στην Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, πω τα μικρά αεροδρομία είναι σε τελείω διαφορετική κατηγορία από το Χίθρο, τη Φραγκφούρτη, του Δουβλίνο. Είναι κάτι το ξεχωριστό που είναι συστατικό στοιχείο της ε, περιφερειακής ανάπτυξης. Και επειδή μίλησε και ο κύριος Μπράντμπεν και οι υπόλοιποι μιλητές για τι μία χειραποσκευή και τα υγρά ε, ζελέ και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κράμερ και ο κύριος Χαντραουή οι μεγάλες εταιρείες ε, κάνουν ό,τι θέλουν με τα μικρότερα αεροδρόμια και τους λένε αν δεν σας αρέσει θα σταματήσουμε να ερχόμαστε εδώ. Οπότε είναι δύσκολο να βρούμε την ισορροπία αφενός δηλαδή μεταξύ Τη ύπαρξη του αεροδρομίου και τη ε, ισχύω ε, των αεροπορικών εταιριών όσον αφορά την ασφάλεια. Έχω καταθέσει μια τροπολογία, μια δική μου και άλλη μια συνεργασία με άλλους συναδέλφους για το ποιο πληρώνει την ασφάλεια στο αεροδρόμιο. Υπάρχει πρόβλημα για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Δεν έχουν τι οικονομίε κλιμακό των μεγαλύτερων αεροδρομίων. Οι προπολογισμοί είναι πάρα πολύ μικροί. Και επειδή βεβαίως έχουν ε, μικρούς αριθμούς ε, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Οπότε θα μπορούσαν να έχουν ένα μεγαλύτερο περιθώριο συμμόρφωσης ε, με τα μέτρα ασφαλείας. Η άποψή μου για το να πληρώνει το κράτος δεν ξέρω, εγώ θεωρώ πως θα έπρεπε να ενσωματώνεται στο κόστος λειτουργίας του αεροδρομίου όπως το duty free και οι λοιποί φόροι και τέλη και τα λοιπά. Ένα πρόβλημα που έχω, έχουμε καταθέσει μια σχετική τροπολογία, την 148, είναι ένα νέο φαινόμενο για ε, τέλη ε, στις πιστοτικές ε, κάρτες ε, επιτόπου πρέπει να σταματήσει αυτό γιατί υπάρχει η λεγόμενη δωρεάν επιλογή πληρωμής αν έχει την πιστοτική κάρτα της εταιρείας και έχουν πολύ υψηλές μηνιαίες χρεώσεις ψηλότερες από τις κανονικές πιστωτικές κάρτες οπότε δεν συμφέρουν τον καταναλωτή και σε σχέση με αυτό το οποίο θα συζητήσουμε αργότερα την έκθεση Taylor έχω καταθέσει μια σχετική τροπολογία. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Μπράντμπον, όπω είπαν όλοι, πράγματι πρέπει να τον συγχαρούμε. Σα ευχαριστώ, κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να επενέσω την εργασία του κυρίου Μπράντμπορν αυτό το κείμενο μέσα στα πλαίσια του πακέτου για τις αεροπορικές υπηρεσίες. Ήταν ένα αναγκαίο κείμενο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπράντμπορν που έλαβε υπόψη της τροπολογής μου 7 και 11. Θα ήθελα να πω ότι στην 7 η 65 η δική μου όπου τίθενται τα θέματα ε, για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης είναι κάτι το πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για απερίμωση ορισμένων αεροδρομίων. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή να μελετήσει την κατάσταση και να δει πώς, αν υπάρχουν καταχρήσεις και δεσπόζουσα θέση. Θα πρέπει λοιπόν να μας πει πώς το αντιμετωπίζει. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στις άλλες τροπολογίες τονίζω την θέση ορισμένων αεροδρομίων γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ε, ροή και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Επιτροπή κάτι θα πρέπει να κάνει για αυτό τον εποχικό χαρακτήρα που υπάρχει σε ορισμένα αεροδρόμια μέσα στα πλαίσια και των χρονοθυρίδων. Γιατί ένα θέμα είναι η διαχείριση των σλότ και των αερογραμμών και ένα άλλο θέμα είναι η χωρητικότητα των περιφερειακών αεροδρομίων που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριος Βόλβεν. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σχολιάσω την έκθεση αυτή. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησα την όλη συζήτηση και να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Μπράντμπορν για το ότι ασχολήθηκε με το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα και ένα ζήτημα τελικά το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα και τα μέλη της Επιτροπής αυτής. Και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι η περιφερειακή προσβασιμότητα βρίσκεται πραγματικά στον πυρήνα των όσων θέλουμε να πετύχουμε στα πλαίσια τη εσωτερική αγορά. Θεωρούμε λοιπόν ότι αποτελεί κεντρικό ζήτημα εργασίας και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πολύ σύντομα να ασχοληθώ με τέσσερα ζητήματα τα οποία ακούσαμε. Και ζητώ συγγνώμη αν επαναλαμβάνομαι κατά κάποιο τρόπο με τις παρατηρήσεις μου αυτές. Όσον αφορά το ζήτημα του ορισμού των περιφερειακών αεροδρομίων, Συμφωνούμε με την γενικότερη πρόθεση που υπάρχει εδώ πέρα, το ότι επιθυμείτε να βρείτε έναν ορισμό προκειμένου να απλουστευτούν τα πράγματα και να είναι σαφές σε όλους τι εννοούμε όταν λέμε «περιφερειακός αερολιμένας». Ωστόσο πιστεύω ότι είναι σαφές ότι ο τομέας αυτός δεν έχει ρυθμιστεί και δεν έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε σε έναν συγκεκριμένο αυστηρό ορισμό. Και μόνο και από τις τροπολογίες που έχουμε μπροστά μας βλέπουμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε έναν ενιαίο ορισμό. Και συνέχεια να το χρησιμοποιήσουμε και για άλλες έννοιες, όπως για παράδειγμα οι χρονοθυρίδες ή τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Σας λέω λοιπόν εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε έναν ενιαίο ορισμό. Και με αυτό συνδέεται και το όλο ζήτημα της περιφέρειας επιπτώσεων των περιφερειακών αεροδρομίων και αν θα πρέπει τελικά τα περιφερειακά αεροδρόμια να διαδραματίσουν ένα σημαντικότερο ρόλο στα πλαίσια του κεντρικού δικτύου των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυτή τη στιγμή ότι μόνο τα βασικά αστικά αεροδρόμια, τα οποία αποτελούν κομβικά αεροδρόμια, αυτά τα οποία έχουμε σε περιοχές όπως οι πρωτεύουσε ή εκεί όπου κατοικούν πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι, ότι αυτά θα πρέπει να ενταχθούν αμέσως στο κεντρικό δίκτυο θεωρούμε ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια δεν αποτελούν κομβικά αεροδρόμια, αλλά συνδέονται με κάποια κομβικά αεροδρόμια. Μπορούν λοιπόν τα περιφερειακά αεροδρόμια να δραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την περιφερειακή προσβασιμότητα. Πρέπει λοιπόν να δυναμώσουμε σαφώς ε, τον ρόλο τους, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχουν. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι οι κρατικές ενισχύσεις γνωρίζετε ότι εμεί θέλουμε να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση στον τομέα αυτό, η οποία να συμφιλιώνει την προώθηση αφενός ενός ολοκληρωμένου δικτύου περιφερειακών αεροδρομίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με, από την άλλη, την δυνατότητα να βρεθεί ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού προκειμένου τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων να δαπανώνται με τρόπο λογικό και να μην έχουμε επικαλύψεις όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν τα περιφερειακά αεροδρόμια. Ο κύριος Αλμούνιο, αρμόδιος επίτροπος, ασχολείται με το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων και την αθεώρηση του συστήματος αυτού και στα πλαίσια των περιφερειακών, της αναθεώρησης συστήματος αυτού θα ασχοληθούμε και με τη χρηματοδότηση των περιφερειακών αεροδρομίων και να αναφερθώ και στο ακαθόδε αυτό ζήτημα της ε, μίας χειραποσκευής. Ακούσαμε πολλές παρατηρήσεις σήμερα το απόγευμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα σε δύο ξεχωριστά κατεμέ ζητήματα. Υπάρχουν κάποια συγκρουόμενα επιχειρησιακά συμφέροντα, καθώς επίσης και συμφέροντα των επιβατών, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των εταιριών. Όταν μιλάμε για πρακτικές που ακολουθούν τα αεροδρόμια, εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ισορροπία προσπαθούμε να πετύχουμε ανάμεσα στους πολιτές λιανικής, τις αεροπορικές εταιρείες και τα περιφερειακά αεροδρόμια. Και θα πρέπει να αποφευχθεί βέβαια κάθε κατάχρηση εξουσίας. Οπουδήποτε προκύπτουν αντικρουόμενα τέτοια ζητήματα ή αντικρουόμενα συμφέροντα, θα πρέπει αυτά επιτόπου να επιληθούν και να μην καταλήξουμε αναγκαστικά σε μια κοινοτική νομοθεσία. Όταν μιλάμε όμως για τις επιπτώσεις μπορεί να έχει ο κανόνας της μία χειραποσκευής για τους επιβάτες, συμφωνούμε με αυτό το οποίο είπατε, ότι πολλές φορές προκαλείται σύγχυση στους επιβάτες από αυτές τις πολλές διαφορετικές πολιτικές που υπάρχουν και που διαφέρουν από τον αεροδρόμιο στο άλλο. Οι συνάδελφοί μου θα μελετήσουν το ζήτημα αυτό, όσον αφορά δηλαδή τις επιτρεπόμενες αποσκευές, στα πλαίσια της μελέτης αντικτύπου για την πιθανή αναθεώρηση του κανονισμού 261. Ξεκίνησε επίση και μια δημόσια διαβούλευση που θα μα επιτρέπει να συλλέξουμε τι απόψει των ενδιαφερομένων μερών για το ζήτημα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να εκφράσω τι απόψει μου και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ το ζήτημα αυτό. Κύριο Μπράτμουν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Απλώς θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σχόλια έτσι ώστε να συγκλίνουν όλες αυτές οι παρατηρήσεις και με βάση αυτά που είπε και η Επιτροπή. Ως προς θέματα ανταγωνισμού έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτή την έκθεση, να εστιάσουμε το θέμα μας στη, στην ίση πρόσβαση όλων των φορέων δεν πρόκειται μόνο για τη μία χειραποσκευή, αν και αυτό είναι σημαντικό, γιατί βεβαίως υπάρχει θέμα ανταγωνισμού και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι αερο, αερομεταφορείς που θέλουν να περιορίσουν τις αποσκευής γιατί θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους εμπλό. Μιλάμε όμως και για υπηρεσίες που ε, προβάλλουν αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια. Για, τα, για το πρόγραμμα TEN, επειδή εγώ ήμουν εισηγητής το 1999 2004 είχαμε ασχοληθεί με αυτά τα κομβικά ε, δίκτυα που θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τα αεροδρόμια και να ενθαρρύνουν τα περιφερειακά αεροδρόμια χωρίς ε, να ε, επιβάλλουν το σκέλος της κρατικής ενίσχυσης. Στα πρώτο πρόγραμμα TENS δεν ελήφθη υπόψη, γι' αυτό το επαναλαμβάνω εδώ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και ότι η Επιτροπή συμφώνησε. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος Χίγγινς, αν είναι εδώ, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, ως προς την ασφάλεια. Αρχικά, Πρόεδρε, ήθελα να κρατήσουμε τη θέση μας ως Κοινοβούλιο. Μόσαστε ότι στις συζητήσεις μας για την αεροπορική ασφάλεια είχαμε ζητήσει πιο αυστηρά μέτρα πέρα από τη γενική ασφάλεια και αυτό προ, προσπάθησα να διατηρήσω εδώ, μέσα στα πλαίσια της αναλογικότητας, δηλαδή της ε, δημόσιας ε, επιδότησης σε σχέση με τον ναύλο. Ο κύριος Πέρκερ μίλησε για το ότι τα περιφερικά αεροδρόμια θα πρέπει να γίνουν πιο δελεαστικά. Δεν μιλάμε για έλλειψη περιορισμών, αλλά τα ίδια, για το ότι τα ίδια αεροδρόμια γίνονται πιο δελεαστικά, ελκυστικά, γιατί είναι πιο ε, φιλικά προς τον καταναλωτή. Προσπαθώ να το αντιμετωπίσω. Ο κύριος Σασόλη, προς τον κύριο Σασόλη έχω να πω τα εξής. Με τις τροπολογίες αυτού, νομίζω ότι αναφέρθηκε στην υπαριθμόν 1, θα ήθελα να τη λάβω υπόψη ε, μέσα στα πλαίσια της πρότασης συμβιβασμού. Ως προς την 39 της κρατικές επιδοτήσεις, αν θέλουμε να κάνουμε διαφοροποίηση της, ε, των χρηματοδοτήσεων αυτών, γιατί μιλήσαμε για δημόσιες υπηρεσίες και ότι είναι ζωτική σημασίας για απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν υπάρχουν άλλες μορφές βιώσιμης μεταφοράς. Υπάρχει και το θέμα της αρχικής βοήθειας, της αρχικής επιδότητας, Startup Aid, εκεί όπου γίνεται, ορίζεται μία νέα διαδρομή και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι βιώσιμη. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν περιορισμοί, διότι δεν θα ήθελα να ξεκινήσει μια υπηρεσία να χρηματοδοτείται και μόλις ε, αρχίσει να πρέπει να περιοριστεί. Ως προς τον κύριο Ούτζες, προς την κυρία Μάισνερ δηλαδή, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που προσπαθώ να δω στις προτάσεις συμβιβασμού. Όπως είπε ο κ. Τέιλορ, έχει μπει το θέμα των ε, ΑΜΕΑ δεν είναι ένα θέμα που αφορά τα περιφερειακά αεροδρόμια, αφορά όλα τα αεροδρόμια. Είτε είναι κανείς στο Χήθρο, είτε σε ένα απομακρυσμένο σκοτικό αεροδρόμιο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνει στα πλαίσια των δικαιωμάτων των επιβατών και όχι να κατακαιρματιστεί. Θα ήθελα να το αναφέρετε στον κύριο Ούτζες. Ο κύριος Κράμερ μίλησε για τη διατροπικότητα, την κρατική, τις κρατικές επιδοτήσεις. Ε, μιλήσαμε και για το ticketing ως προς τη διατροπικότητα. Και τέλος, ο, οι κύριοι Higgins και Ελ Καντράουι μίλησαν για διαφάνεια των ε, ε, ναύλων. Δεν θα πρέπει να είμαστε απαγορευτικοί. Θα πρέπει όπως είπα και αρχικά, να δούμε κατά πόσο υπάρχουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις να είναι διαφάνειας, δηλαδή οι πολίτες να λαμβάνουν αυτό για το οποίο καταβάλουν το αντίτιμο. Ε, αν χρησιμοποιούνται λοιπόν χρεωστικές ή πιστοτικές κάρτες θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να καλύπτεται το συνολικό κόστος και να μην υπάρχουν συμπληρωματικές ε, χρεώσεις που να μην είναι διαφανείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε κυρία Μπράτμπορν. Η Επιτροπή θα γίνει στις 27 Μαρτίου και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια στην πρώτη σύνοδο του Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ. Δικαιώματα των πολιτών, ο κύριος Τέιλορ. Επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρος, έχουμε μία ώρα για το ζήτημα αυτό, Κίθα. Θα προσπαθήσω να μην αναλώσω όλη αυτή την ώρα, λέει ο κύριος Τέιλορ. Να ευχαριστήσω καταρχάς του σκιώδης εισηγητής εισηγητές με συγχωρείτε, οι οποίοι με βοήθησαν να καταρτήσω την έκθεση αυτή. 195 τροπολογίες συνολικά υπευλήθησαν, συν 30 παράγραφοι, νέοι παράγραφοι, από την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Από τις 195 αυτές τροπολογίες καταλήξαμε σε 13 συμβιβαστικές τροπολογίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν περίπου 60 ε, από τις αρχικές τροπολογίες, καλύπτουν 60 και παραπάνω από τις αρχικές τροπολογίες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια πολύ καλή συνένεση για την έκθεση αυτή αύριο. Εξ αρχής είχα πει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη νομική διαφάνεια και μία ομοιόμορφη εφαρμογή όσον αφορά τους κανονισμούς για τα δικαιώματα των, ατόμων που ταξιδεύουν αεροπορικά σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην ξεχνάμε ότι η έκθεση αυτή έχει να κάνει με τα δικαιώματα των επιβατών. Προσπάθησα να καλύψω πολλά ζητήματα διεξοδικά στην έκθεση αυτή, την αναθεώρηση του κανονισμού 261 και του κανονισμού 11.07 καλύπτοντας ε, και τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρίες και των ανθρώπων περιορισμένης κινητικότητας. Επίσης η έκθεση αυτή κάνει κάποιες γενικότερες συστάσεις. Κάποια βασικά σημεία της έκθεσης αυτής στα πλαίσια του γενικότερου αυτού πλαισίου είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια η οποία απαιτείται όσον αφορά τις τιμές Ακούσαμε ήδη πολλές φορές σήμερα το απόγευμα να γίνεται λόγος για το ζήτημα αυτό, το ότι πρέπει να αντικατοπτρίζει η προτινόμενη τιμή ενό εισιτηρίου την πραγματική τιμή που τελικά καταλήγει να πληρώνει ο επιβάτης. Επίσης, ε, χρηματοοικονομική προστασία των επιβατών αν χαροκοπήσει μια αεροπορική εταιρεία. Και θα πρέπει η αεροπορική αυτή εταιρεία να παρέχει άμεσα ενισχύσεις προς επιβάτες σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο και αν δραστηριοποιείται. Και θα πρέπει να εξηγείται επίσης και στους ε, επιβάτες ποιο είναι ο περιβαλλοντικό αντίκτυπος των ε, ταξιδιών που κάνουμε με το αεροπλάνο. Αν επιθυμούμε πραγματικά να μειώσουμε τα τις εκπομπές ε, του θερμοκηπίου, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει και ο πελάτης και ο επιβάτης πώς επηρεάζει το μέσο το οποίο έχει επιλέξει το περιβάλλον. Επίσης, ε, ζητάμε μία τη δημιουργία ανεξάρτητων αυτόνομων φορέων επιβολής ε, της νομοθεσίας, ομοιόμορφα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα τον κανονισμό 261 και σας υπόσχομαι να μην μακρηγορήσω κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά λοιπόν τον κανονισμό 261 ζητάμε σχετικά με αυτόν να έχουμε σαφή πληροφόρηση και προσβάσιμες πληροφορίες. Δηλαδή, ο επιβάτης να μπορεί σε κάθε φάση της κράτησης αλλά και του ταξιδιού να μπορεί να έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Θέλουμε επίσης να υπάρχουν αποσαφηνήσεις σε οποιονδήποτε νέο κανονισμό για συγκεκριμένους ορισμούς, ιδίως όσον αφορά τις έκτακτες περιστάσεις και όσον αφορά την ακύρωση της πτήσης. Επίσης λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια αντιμετώπισης των κατακυλιών των παραπώνων των επιβατών τόσο από την αεροπορική εταιρεία όσο και από τα όργανα επιβολής νομοθεσίας. Και όσον αφορά τώρα τον κανονισμό 1107 για τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, εδώ ζητούμε μία πρόσβαση χωρίς εμπόδια στα αεροδρόμια και στα αεροσκάφη. Ζητάμε ιατρικό οξυγόνο να είναι διαθέσιμο μέσα στο αεροπλάνο, μέσα στο αεροσκάφος και ζητάμε και υψηλότερα επίπεδα υποβοήθησης για τους ανθρώπους αυτούς προκειμένου να μπορούν να έχουν μια εξασφαλισμένη θέση μέσα στο αεροσκάφος. Επίσης ζητάμε να υπάρχει και μία αποζημίωση όσον αφορά τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτοί όσον αφορά τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με περιορισμένη κινητικότητα ή με αναπηρία. Η αποζημίωση προβλέπεται αυτή τη στιγμή καλύπτει μόνο κάποιε εκατοντάδε ευρώ, ενώ πολλέ φορέ ο εξοπλισμό που χρησιμοποιούν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και κοστίζει χιλιάδε ευρώ. Όσον αφορά τώρα τη συμβαστική τροπολογία Β. Στην προηγούμενη συνεδρίαση που είχαμε του σκιώδεις συζητητέ συζητήσαμε τις, το ζήτημα των συμβουλευτικών ομάδων όσον αφορά τους επιβάτες και όσον αφορά την αποζημίωση των επιβατών όταν καταπατώνται τα δικαιώματά τους. Θεωρήσαμε λοιπόν θα πρέπει να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνουν οι συμβουλευτικές αυτές ομάδες, ποιος είναι ο ρόλος τους. Δεν θα δώσω αυτή τη στιγμή όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης γίνεται μία αναφορά και σε άλλες δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Υπάρχει μία διαθέσιμη ιστοσελίδα καθώς επίσης και κάποιες εθνικές εκστρατείες. Και γίνεται και μία αναφορά και σε μία εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα νέα ευθύ κινητά και η οποία είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή αυτή λοιπόν θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και σχετίζεται και με τη συμβαστική τροπολογία Γ, η οποία ζητεί παροχή πληροφοριών σε περισσότερες γλώσσες. Εν κατακλείδη, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους κοιόδης ηγητές και τη γραμματεία για την υποστήριξή τους και ελπίζω ότι το θετικό αυτό πνεύμα συνεργασίας θα φανεί και σε μία θετική υπερψήφιση της έκθεσης αύριο. Σας ευχαριστούμε κύριε Τέιλερ, ο κύριος Σασόλη για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τέιλορ για την δύσκολη αυτή εργασία και γιατί ε, δείχνει πνεύμα συνεργασίας στις υποδείξεις μας ως προς τις προτάσεις συμβιβασμού όπως συνηθίζεται, όπως ισχύει, δεν είναι ικανοποιητικές για όλους κατά 100% αλλά συγκλίνουν προς μία κατεύθυνση. Και σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μεμονωμένες διατάξεις του εγγράφου. Κατά την εργασία μας προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη το θέμα της καλύτερης πληροφόρησης ως προς τα δικαιώματα των επιβατών. Το έγγραφο τονίζει αυτή την ανάγκη σε πολλά σημεία και μιλά για άμεση επαφή μεταξύ των επιβατών και των αερομεταφορέων καθώς και, τις, ε, και συγκεκριμένες διατάξεις και προδιαγραφές ε, με βάση πληροφορίες στην ιστοσελίδα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αθέμητες, να ενθαρρύνονται αθέμητες πρακτικές δηλαδή όταν η αρχική τιμή διαφέρει από την τελική ή ορισμένα μη δικαιολογημένα έξοδα. Το, ο, ο επιβάτης θα πρέπει να μπορεί να διορθώσει κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια της κράτησης. Δηλαδή όταν ένα γράμμα δεν έχει γραφτεί σωστά, δεν έχει αναγραφεί σωστά. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση στην Πολωνία. Δηλαδή το επίθετο μιας γυναίκας διαφέρει κατά ένα γράμμα από το επίθετο του άνδρα. Και εάν γίνει αυτό το λάθος, αυτό το ένα γραμματάκι μπορεί να σημαίνει πολύ υψηλό αντίτιμο. Επίσης, ο επιβάτης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποσύρει την κράτηση μέσα σε δύο ώρες. Γιατί υπάρχουν ορισμένες πρακτικές που θα πρέπει να αποθαρρύνουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε προσφορές, δηλαδή 100 ευρώ αναπτύσσει, αλλά όταν υπολογιστεί η τελική τιμή φτάνουμε σε 200 ευρώ. Άρα δεν πρόκειται για χαμηλή τιμή, για μια καλή προσφορά ή για την καλύτερη δυνατή. Κατανοώ ότι ο εισηγητής θέλει μεγαλύτερη χρονική περίοδο, αλλά νομίζω ότι δύο ώρες είναι αρκετές για να φτάσουμε στο συμπεράσμα ότι ε, έχουμε κάνει ένα λάθος και θέλουμε να αποσυρθούμε να αποσύρουμε την κράτηση. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή και μπορώ να πω ότι εξεπλάγει από τα λόμπι γιατί λάβαμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από ένα συγκεκριμένο λόμπι που εκπροσωπεί αερομεταφορείς. Λένε ότι τα μικρά παιδιά που ταξιδεύουν τα παιδιά δεν είναι PRM. Αν όχι αυτοί, τότε ποιοι. Έχουμε όμως ε, διάφορες κατηγορίες. Μιλάμε δηλαδή για πρόσωπα με περιορισμένη κινητικότητα ή για άλλες αναπηρίες. Γιατί έχει σημασία να μιλάμε για γονείς και γονείς που συνοδεύουν μικρά παιδιά. Με εκπλήσει η ε, στάση των αερομεταφορέων γιατί τα αεροδρόμια βοηθούν τα πρόσωπα με περιορισμένη κινητικότητα. Δεν το κάνουν οι αερομεταφορές. Όπως λέει και το κείμενο όπως λέει και το κείμενο, θα πρέπει ο κύριος Σταγιάννη να αποφανθεί επί του θέματος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο νομοθέτης ήθελε να νομοθετήσει όχι μόνο για τα αμαία, αλλά για μια ευρύτερη κατηγορία, η οποία ονομάζεται PRM, δηλαδή πρόσωπα με περιορισμένη κινητικότητα. Γι' αυτό ο τίτλος μιλά για δικαιώματα προσώπων με περιορισμένη κινητικότητα μεταξύ άλλων. Συνεπώς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι εφόσον το άρθρο 2 του κανονισμού ε, αναφέρεται σε προβλήματα λόγω ηλικίας, τα παιδιά θα πρέπει να θεωρούνται PRM τη στιγμή που δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δημόσιες μεταφορές θα πρέπει να, συνοψίσ, να συνοψίσετε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε ένα λεπτό παραπάνω. Κύριο Σασόλη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα οι συγητές έχουν μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Τέιλορ, για αυτή την εργασία σε, αυτό το, σε αυτή τη φάση των τροπολογιών συμβιβασμών. Νομίζω ότι συνολικά είναι πολύ καλή η εργασία. Έχουν μπει τα βασικά θέματα που έχουν φυγεί από τις τροπολογίες. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω διότι έλαβε υπόψη τη δική μου πρόταση σε σχέση με το αντίτιμο που καταβάλλεται για τα μικρά παιδιά, τα ανήλικα. γιατί σε αυτή τη φάση που διανύουμε, τη φάση κρίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά. Θα ήθελα να κάνω μόνο δύο παρατηρήσεις σε σχέση με το συμβασμό H. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η κυρία Αγιάλα Σέντερ Μιλά για τη δυνατότητα που θα πρέπει να έχουν οι επιβάτες που ταξιδεύουν με μικρά παιδιά να έχουν προτεραιότητα κατά την επιβίβαση αλλά θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα πρόσωπα περιορισμένης κινητικότητας. Θα ήθελα ο κύριος Τέιλορ να δεχτεί και μία προφορική τροπολογή από την κυρία Σεναλόβα σε σχέση με τα δικαιώματα των επιβατών κατά τη στιγμή της κράτησης του εισιτηρίου. Κύριε Τέιλορ, αυτό θα μπορούσε να ε, εισαχθεί στην πρόταση συμβασμού C. Πρόκειται για τις ε, πλήρεις πληροφορίες ως προς τα δικαιώματα των επιβατών και την, την επικοινωνία, με συγχωρείτε, τη γλώσσα επικοινωνίας κατά την κράτηση του εισιτηρίου. Η τροπολογία συμβασμού Γ θα μπορούσε να έχει ως εξής και σας διαβάζω. Υπογραμμίζει ότι οι πλήρεις πληροφορίες για τα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να κοινοποιηθούν είτε από τους ε, αερομεταφορείς είτε από τους tour operators ε, στη γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά την κράτηση του εισιτηρίου. Και μετά το κείμενο ως έχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Γκρίσμπεκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Τέιλορ για την έκθεσή του και για τις πολύ καλές σχέσεις μας ε, με καλό πνεύμα συνεργασίας, χιούμορ και ούτω καθεξής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τροπολογίες συμβιβασμού επέτρεψαν όχι τη συνένεση 100%, αυτό θα ήταν και ανησυχητικό μπορώ να πω, αλλά να προσεγγίσουμε τις θέσεις μας εξαιτίας της αμοιβαία εργασίας, σύγκλησης απόψεων, ιδιαίτερα ως προς τη διαφάνεια, την πληροφόρηση, τα στοιχεία διευκρίνησης που χρειάστηκαν και χαίρομαι για το περιεχόμενο των προτάσεων συμβασμού. Είχαμε 195 τροπολογίες αρχικά, συν ε, τις τροπολογίες συμβιβασμού. Βλέπουμε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η έκθεση για τα δικαιώματα των επιβατών και τα δικαιώματα των πολιτών ως προς την κινητικότητα και βλέπουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να συγκεκριμενοποιεί αρκετά θέματα. Ορισμένες επιφυλάξεις τώρα θα ήθελα να εκφράσω. Ως προς το συμβασμό H, δηλαδή τις οικογένειες που ταξιδεύουν με μικρά παιδιά, χωρίς να επηρεαστούμε από τους αερομεταφορείς, αναρωτιέμαι κατά πόσο δεν πάμε κάπως μακριά. Βεβαίως θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις οικογένειες που ταξιδεύουν με μικρά παιδιά. Επειδή και εγώ ε, είχα πολύ μικρά παιδιά, μικρά παιδιά και χρειάστηκε να ταξιδέψω με αυτά. Ιδιαίτερα η κατά προτεραιότητα επιβίβαση να χρησιμοποιούνται τα καροτσάκια μέχρι την, την επιβίβαση, το σημείο επιβίβασης. Επίσης να εγκαταλείπουν το αεροσκάφος κατά προτεραιότητα. αλλά επίσης και οι οικογένειες θα πρέπει να συνδράμουν, να είναι συνεργάσιμες. δεν θα πρέπει να θεωρούνται πρόσωπα περιορισμένης κινητικότητας. Δεν μπορούμε να τους εξομοιώσουμε με αυτή την κατηγορία γιατί αποδυναμώνει την ε, έννοια του ε, PMR. Γι' αυτό στην τμηματική ψηφοφορία θα εκφράσουμε επιφύλαξη αύριο, το πρωί δηλαδή, που θα ψηφίσουμε ως προς τη συμβουλευτική ομάδα, ως προς τη, τα δικαιώματα των επιβατών. Ευχαριστώ τον κύριο Τέιλορ γιατί έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο διάλογο. Ε, όχι σε συνθήκες κρίσης, αλλά γενικότερα θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση. Ευχαριστώ για, αυτό το, για αυτές τις διευκρινήσεις. Ως προς τα ε, στοιχεία, προσωπικά στοιχεία επιβατών, PNR, χαίρομαι διότι οι επιβάτες πληροφορούνται για το περιεχόμενο των στοιχείων που ε, κατακρατούν οι αρχές και τη νομική ασφάλεια που υπάρχει σε σχέση με το PNR. Ε, Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση της μη πρόσβασης ενός επιβάτη. Στο ΚΑΠΑ, στο συμβιβασμό, μιλάμε για αποζημιώσεις για απολεσθέντα ε, πάνω από 6 ώρες. Σας ευχαριστώ πολύ και θα δεχτούμε τις περισσότερες τροπολογίες συμβιβασμού. Ευχαριστώ κύριε Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Είχαμε ενδιαφέρουσες συναντήσεις και πριν από κάτι εβδομάδε όταν προσπαθήσαμε να βρούμε συμβιβασμούς, ε, κάποιους συμβιβασμούς, οπωσδήποτε μπορούμε να τους υποστηρίξουμε, αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ε, δεν μπορούμε. Σύντομα θα τους διατρέξω. Αρκεί να πούμε πως το όλο ζήτημα του γιατί κοιτάμε αυτό το θέμα, που δεν το τονίζουμε αρκετά, είναι γιατί υπήρχε ένα ζήτημα που λεγόταν ε, φεστιακή τέφρα. Καταστροφικό και πρωτόγνωρο. Ο άλλος λόγος ήταν οι αποφάσεις του ΔΕΚ και δεν ακούσαμε τίποτα από την Κομισιόν σχετικό, αν μου επιτρέπετε. Μια αναφορά παρόδο. Αλλά, σύντομα, κύριε Πρόεδρε, να πω το εξής για την ε, συμβαστική λύση ε, τροπολογία Α. Το πρώτο μισό οπωσδήποτε το υποστηρίζουμε. Το δεύτερο μέρος ε, δεν ξέρω, επαναλαμβάνεται και γίνεται και δύσκολο, πολύπλοκο. Και έχουμε κάποια δυσκολία μετά τη λέξη Ευρώπη για τη συμβουλευτική ομάδα τώρα. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις πληροφορίες γιατί δεν ξέραμε ποια ήταν τα μέλη αυτής της ομάδας για τη συμβαστική ΣΥ και εδώ παρέχουμε κάποια ερωτήματα γιατί είναι πολύπλοκο, γιατί μιλάει για σημεία κλειδιά του ταξιδιού. Ναι, εντάξει, να έχουμε καλή επικοινωνία. Έχουμε όμως πρόβλημα με την διατύπωση. Η αρχή δεν είναι ε, λανθασμένη για την ε, συμβαστική δέλτα. Οπωσδήποτε, ναι, παρουσία ανθρώπων και τα λοιπά στα αεροδρόμια, αλλά έθεσα πάλι το ζήτημα της ε, επιστροφής των χρημάτων απευθείας. Ε, στο αεροδρόμιο. Αλλά δεν θα εμφανιστεί βεβαίω το προσωπικό εδάφος με μια βαλίτσα μετρητά. Οπότε, ναι, βοηθή, ναι, εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτή τη λέξη. Η ε μετά. Το PNR το έχουμε κουράσει πια εδώ και χρόνια. Αν θέλετε πως πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ πέρα, εντάξει, εμείς δεν το θεωρούμε, αλλά... Σίγμα ταφ, για τη διαφάνεια των τιμών συμφωνούμε. Πράγματι δεν μπορεί κάποιο να μπαίνει στο ίντερνετ, να φτάνει ένα ειστήριο και μέχρι να φτάσει στην τελευταία σελίδα, τέσσερι σελίδε μετά, να έχει τριπλασιαστεί η τιμή. Οι καλέ εταιρείε φροντίζουν να γνωστοποιούν την ε, τιμή στη δεύτερη σελίδα. Αυτή είναι καλή επικοινωνία. Ζήτα. Ναι, Πράγματι το υποστηρίζουμε. Τώρα δύο ώρες για ένα ορθογραφικό λάθος. Ο κύριος ε, Σασάδας, πάμε, ο συνάδελφός μας, έχει δύσκολο όνομα. Μπορεί κανείς να το μπερδέψει. Αλλά για να φύγει μετά κανείς από την ε, κράτηση δεν ξέρω αν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Τμήμα του συμβιβασμού ναι και μετά πάλι όταν φτάνουμε στα PRM. Αντιλαμβάνομαι τη θέση του συναδέλφου αλλά το PRM είναι αυτό που είναι και το βρέφος ε, είναι βρέφος, δεν είναι άτομο με περιορισμένη κινητικότητα. Ε, οι καλές εταιρείε φροντίζουν να μπαίνουν ε, νωρίς οι οικογένειες όπως και τα άτομα με καροτσάκια. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορείτε να τα γράφετε αυτά τα πράγματα. Και βεβαίω είναι μια εμπορική απόφαση. Αν μια εταιρεία θέλει να το κάνει, μπορεί να το κάνει. Δεν αγκεί να νομοθετούμε για τα πάντα. Συμβαστική ΙΟΤΑ. Δεν ξέρω αν είναι δουλειά της Κομισιόν να ορίζει ποιες είναι οι εξαιρετικές συνθήκες. Είναι ε, διεθνώς αναγνωρισμένες και σε αυτά συμμορφώνονται επιχειρήσεις. Εμείς μπορούμε να το, μιλά, το συζητάμε όλη μέρα, αλλά υπάρχει ήδη μια, ένας διεθνής ορισμός. Ε, συμβαστική J, μια χαρά. Πρέπει να υπάρχουν πράγματι επαρκείς πληροφορίες για όλους τους επιβάτες και μετά υπάρχει το ζήτημα των αποσκευών και της συνθήκης του Μοντρεάλ. Και εδώ πέρα είναι ένα μικρό πρόβλημα γιατί ε, κάποιες εταιρείες σου δίνουν ε, χρήματα αμέσω μετά από λίγες ώρες, άλλες περιμένουν την ασφάλεια. Δεν είναι τόσο απλό. Αλλά πρέπει να τους βοηθούν τους επιβάτες στο στομότερο δυνατόν. Για την ΕΛ. Ναι, συμφωνώ. Πράγματι πρέπει να απαντούν σύντομα στις ε, διαμαρτυρίες και να ενημερώνονται οι επιβάτες. Εγώ θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρχει μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για τα παράπονα των επιβατών γιατί δεν βλέπω γιατί πρέπει να πληρώνει και κανείς για να λάβει μια απάντηση. Αυτό είναι θέμα όμως ξέτησης των πελατών. Δύο τελευταία σημεία. Τέλος, ε, συμβαστική εν, κύριε Πρόεδρε, η τελευταία οπωσδήποτε έχουμε ένα ζήτημα για την ε, βοήθεια του εαυτού του, το τι μπορεί να κάνει κανείς για να βοηθήσει αυτόν. Όχι, αν αγοράσει κανείς εισιτήριο είναι υποχρέωση της εταιρεία μετά να αλλάξει το δρομολόγιο. Το κάνουν οι καλές εταιρείε. Δεν υποστηρίζουμε το να βρει ο καθένας τον τρόπο μόνος του. Αυτά σας ευχαριστώ για την υπομονή σας κύριε Πρόεδρε και ελπίζω ο εισηγητής να βρει και τα σχόλιά μου επικοδομητικά. Μάλιστα έχουμε ακόμα 8 ομιλητές και λιγότερο από 25 λεπτά. Τρία λεπτά λοιπόν για τον κάθε βουλευτή. Ξεκινάμε τον κύριο Μπαχ λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Θέλω να τονίσω δύο ζητήματα. Να συγχαρώ βεβαίω τον κύριο Τέιλορ. Θεωρώ πως στην περίπτωση χρεοκοπίας της εταιρεία θα πρέπει, γιατί είδαμε τις περιπτώσεις Spanair, Malev και λοιπόν ε, εταιριών, ε, μην ξεχνάτε ότι τα τελευταία 10 χρόνια επηρεάστηκαν 2 εκατομμύρια επιβάτες από τέτοιες χρεοκοπίες και θέλω να παραπέμψω εδώ πέρα στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Νοεμβρίου 2009 που προτείνει διάφορες λύσει. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που μου φαίνεται σημαντικό είναι ένα κοινό πλαίσιο πέρα από την έκθεση του συνάδελφου Τέιλορ για τους επιβάτες σε όλα τα μέσα μεταφοράς και οπωσδήποτε πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές και να λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά του κάθε μέσου μεταφοράς αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές και μία συγκρισιμότητα. Και βεβαίως ε, αυτή η ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίου με διαφορετικά μέσα είναι πάρα πολύ σημαντική και παρόλα αυτά θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στο να μην ε, οδηγηθούμε σε χειροτέρευση της ε, κατάστασης και να οδηγηθούμε στον ελάχιστο κοινό παρνομαστή, αλλά να έχουμε φιλόδοξους στόχους. Και νομίζω σε αυτό συνεισφέρει αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριο Αλχαντραουή για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι εξαιρετική η έκθεση που αντιμετωπίζει τα σημαντικότερα πράγματα. Θα περιοριστώ σε δύο σημεία. Πρώτον, ένα σημείο το οποίο ακούστηκε ήδη πάρα πολλές φορές για τη συμβαστική λύση AIDS. Πρέπει να διευκρινίσουμε το τι θα γίνει βεβαίως με την καλύτερη αντιμετώπιση των ε, παιδιών και βεβαίως τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα αλλά όπως είπε και ο κύριος ε, Σασόλη, πράγματι πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην επιβίβαση και να μπορούν να υπάρχουν ε, συνεννοήσεις για το τι θα γίνει με τα παιδικά καρότσια. Όπως είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ που θέλει να μπει στο κείμενο. Πράγματι πρέπει να το πούμε ρητός. Και δεύτερον και κρίσιμης σημασίας να λάβουμε μέτρα για την ε, ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε καλύτερα τον αντίκτυπό τους. Και αυτό συγκεκριμένα σημαίνει πως οι εθνικοί οργανισμοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση για να αντιμετωπίζουν τις ίδιες καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο. Ένα δίκτυο λοιπόν των εθνικών αρμοδίων αργών είναι ένα σημαντικό βήμα και θα μπορέσουμε μετά να κάνουμε μια καλύτερη ε, χρησιμοποίηση στατιστικής ανάλυσης και χρήσης των στοιχείων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης μεταξύ κρατών και εταιριών. Και για μελλοντικά μέτρα το ίδιο. Οπότε αυτό νομίζω γίνεται και στην παράγραφο 2 και στην 3α και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε λιγότερο χρόνο από 3 λεπτά Ήδη ο αριθμός των σχολείων δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση, συμπληρώνει το πακέτο των αεροδρομίων και ευχαριστούμε τον εισηγητή. Όλοι έχουμε τις εμπειρίες μας με τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών, τη μη τους. Ε, σε τρία σημεία θα αναφερθώ σύντομα. Σημαντική είναι η διαφάνεια και χρειάζεται πρόσβαση σε πληροφορίες. Αυτό είναι κάτι στο οποίο υπάρχει πραγματικά έλλειμμα και θα πρέπει σε περίπτωση επίσης χρεοκοπίας να υπάρχει δυνατότητα βοήθειας των επιβατών. Στη Sky Europe νομίζω υπήρξε κάποια παρέμβαση και τρίτον και το ανέφεραν αλλά θέλω και εγώ να το τονίσω κάποιοι συνάδελφοι για την κυρία Σασάδα. Ε, τα παιδιά δεν είναι ανάπηροι. Εντάξει, βεβαίως γίνονται, υπάρχουν οι προβλέψεις για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και εποφελούνται από αυτό και τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, αλλά δεν πρέπει να ανακατεύουμε τους όρους. Καλύτερο είναι νομίζω να, να παραμείνουμε σε μια διάκριση αυτών των πραγμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ για τρία λεπτά. Ναι, και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή. Στην παράγραφο 22 αναφέρεται πως τα δικαιώματα στις καθυστερήσεις θα πρέπει να ισχύουν σε όλα τα μέσα μεταφοράς και λέω, βλέπω εδώ πέρα πως οι δύο μεγάλες ομάδες θέλουν να διαγραφεί. Μιλάμε για δίκαιο ανταγωνισμό. Ε, πώς εξηγείται αυτό. Εγώ ταξίδεψα προσφάτως από το Βελιγράδι στη Βιέννη, ε, χιόνιζε στη Βιέννη, έξι ώρες καθυστέρηση, δεν παραπονέθηκα και ήθελαν να μου δώσουν ε, 25 ευρώ. Δεν τα πήρα. Αλλά βλέπετε τι γίνεται. Όταν καθυστερήσει ο σιδηρόδρομος, περνάει ο ελεγκτής, μοιράζει τα κουπόνια γιατί είναι ο νόμος, συμμορφώνονται και τελειώνει. Στο αεροδρόμιο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάπου να απευθυνθούς. Υπάρχει τώρα ένα ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο, το EU Claim λέγεται. Απευθύνθηκα σε αυτού. και τι κάνουν. Αυτοί έχουν το μοντέλο το αμερικανικό ότι αν χάσω δεν ε, μου ζητάνε λεφτά, αν κερδίσω κρατάνε 20%. Και τι γίνεται τώρα, πάνε στα δικαστήρια, η Air Berlin, η αεροπορική εταιρεία, καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην εκδοθεί απόφαση. Γιατί ε, αποφάσισε ε, η Κομισιόν πως σε πέντε ώρες ε, καθυστέρηση υπάρχει αποζημίωση στα τρένα μετά από μία ώρα και το ΔΕΚ είπε μετά από τρεις ώρες. Γιατί λοιπόν δεν υπήρξε τελικά κάποια απόφαση για το γιατί να εξαιρεθούν τα αεροπλάνα, τελικά συμβιβάστηκαν με 250 ευρώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Δεν είναι σωστή αυτή η κατάσταση. Και εδώ πέρα απευθύνομαι στι μεγάλε κοινοβουλευτικέ ομάδε. Γιατί είστε κατά αυτού του πράγματο. ίδια δικαιώματα για όλου. Καθυστέρηση έχουμε. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο ανεξάρτητο να επιλύσει το ζήτημα, έχουμε διακριτική μεταχείριση δεν αντιλαμβάνουμε γιατί είστε κατά. Σας παρακαλώ λοιπόν αύριο να υπερψηφίσετε την τροπολογία, να μην διαγραφεί αυτό το σημείο, να έχουν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι επιβάτες ίδια δικαιώματα και να απευθύνονται στην ίδια υπηρεσία. Ευχαριστώ κύριε Σίγκινς. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Τέιλορ, Νομίζω ότι η έκθεση αυτή αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου και υποστηρίζει πραγματικά τα δικαιώματα των επιβατών. 195 τροπολογίες συνολικά. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση μέσω συμβαστικών τροπολογιών. Εμείς 10 ε, τροπολογίες από το ΕΛΚΑ έχουμε συνυπογράψει, οι οποίες ε, θεωρούμε ότι είναι λογικές Προσπαθούμε ουσιαστικά να τακτοποιήσουμε κάπως την έκθεση αυτή και να την κάνουμε λίγο πιο εύχρηστη στην εφαρμογή της. Όσον αφορά την 162, ζητάμε εδώ πέρα μία διαγραφή. Λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ομοιόμορφη ημερομηνία κατά την οποία θα μπορούν οι επιβάτες ε, να αποζημιώνονται. Θεωρούμε ότι στην πράξη όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο σε ε, υπαίθριες περιοχές, σε απομακρυσμένες περιοχές. Ξέρετε ότι οι μεταφορές γίνονται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα. Οι ε, μεταφορές αυτές ε, είναι πολλές φορές πολύ αποτελεσματικές, θεωρώ ότι δεν μπορούμε εκεί πέρα να επιβάλλουμε ομοιόμορφα τα όσα προτείνουμε μέσω της έκθεσης. Γι' αυτό το λόγο κάνω και μια σχετική τροπολογία. Όσον αφορά τώρα την ε, τροπολογία 84, η κυρία Φώστερα αναφέρθηκε σε αυτήν, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν λάθη τα οποία γίνονται κατά, την κράτηση. Εμείς προτείνουμε να μην διορθώνται μόνο τα λάθη κατά την κράτηση, αλλά λάθη online που γίνονται κατά την κράτηση, δηλαδή όταν η κράτηση γίνεται μέσω του διαδικτύου και σε σχέση με τα δεδομένα P ναρ λέμε εδώ πέρα free of charge δωρεάν και η κυρία Φώστρα αναφέρθηκε σε αυτό. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες τροπολογίες, αυτά, αυτά ήθελα να πω κυρίως. Θα αναφερθούμε βέβαια εκ νέου στις τροπολογίες αυτές την ημέρα της ψηφοφορία, πάντως γενικά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τέλειρο για την εργασία που έκανε, κυρία Σαναλόβα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους Κιώδης, όπως έκαναν και οι άλλοι, ιδιαίτερα για τη στροπολογία συμβιβασμού και το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες, σε αρκετές γλώσσες να έχουμε πληροφόρηση δηλαδή στη γλώσσα κράτησης του εισιτηρίου. Ως προς την ε, πτώχευση, η διαδικασία ε, όπως είπαν οι Μπαχ και Μάισνερ, έχω υποβάλει ορισμένες τροπολογίες. Ήδη το 2009 ζητήσαμε από την Επιτροπή να είναι πιο δραστήρια. Και να δούμε ποια θα ε, είναι η αποζημίωση που θα δοθεί σε περίπτωση πτώχευσης μέσα στα πλαίσια της ε, υποχρεωτικής ασφάλισης και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι δεχτήκατε την τροπολογία μας 121 όταν ζητήσαμε από την Επιτροπή να φτάσει σε ένα λεπτομερές ε, ε, κείμενο σε σχέση με τις έκτακτες συνθήκες που αποτελούν πρόσκομα στην πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων. Πολύ αργά μου είπατε. Όχι, λέει ο κύριος Κόλιτσεκ, ε, ε, όποτε το έκανε ο κύριος Φώστερ, το έκανα και εγώ. Ε, τον συμπεριλάβατε αυτόν, εμένα όχι. Όχι, όχι, το αμφισβητώ, λέει ο Πρόεδρος. Άλλη φορά να σηκώνετε το χέρι σαφέστερα. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι καλύτερη από την προηγούμενη και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τέιλορ. Οι τροπολογίες συμβιβασμού είναι αρκετά περίπλοκες και θα τις υποστηρίξουμε κατ' εξαίρεση. Θα πρέπει να έχουμε ε, σαφέστατη τιμολόγηση. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ μικρών παιδιών κάτω από δύο και μεταξύ 2 και έξι. Έχω τέσσερα παιδιά και ξέρω πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Ως προς τα πρόσωπα με περιορισμένη κινητικότητα θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εξοπλισμού και πάνω στο αεροπλάνο έτσι ώστε να μπορούν να μετακινούνται. Ως προς την ε, χρονική περίοδο για αλλαγές κράτησης. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Μερικοί συνάδελφοι είπαν ότι ίσως υπάρχει, υπάρχουν ορθογραφικά λάθη κατά την κράτηση. Τι σημαίνει ελάσσον αλλαγή. Ως προς θέματα ανωτέρας βίας, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται το θέμα να οριστεί εκ νέου για την αποζημίωση στα αεροδρόμια. Δεν χρειάζεται να μεταφέρονται ε, αποσκευές ε, γεμάτες χρήματα. Ε, μπορεί να δοθεί αποζημίωση και στα αεροδρόμια. Συνολικά είναι πολύ καλή έκθεση. Mm, sí, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Τέιλορ για την εργασία του και γιατί έφτασε σε συμβιβασμού σε όλους τους τομείς κατά το δυνατό. Νομίζω ότι θα πρέπει πράγματι να διαφοροποιήσουμε τις οικογένειες με τα παιδιά, παιδιά νήπια δηλαδή, κάτω από δύο ετών ή άνω των ε, δύο. Ε, δυστυχώς όμως έχουμε και προβλήματα υπογεννητικότητας, γι' αυτό αυτοί που κάνουν παιδιά, ε, ας τους διευκολύνουμε τουλάχιστον. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας ορισμός και να μιλάμε για νήπια ε, κάτω το των 2 και μεταξύ 2 και 6. Αυτό αποτελεί προστιθέμενη αξία και ε, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση, ας το πούμε. Οι 141 και 143 σε αυτές τις δύο, ο κύριος Τέιλερ λέει ότι δεν θα τις υποστηρίξει. Στην 143 το καταλαβαίνω, αλλά για την 141 ε, μιλάμε για παράπονα, για διάκριση και για κακή μεταχείριση. Εδώ ε, μιλώ και για μαρτυρίες, ιδιαίτερα για τις εταιρείες χαμηλού κόστους, που υπάρχει κακομεταχείριση, δηλαδή ε, φυσική κακομεταχείριση, για να το πω έτσι. Θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα ιδιαίτερα. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των αποζημιώσεων. Δηλαδή, να μην περιμένουμε την αναθεώρηση όλου του κανονισμού, να πρόκειται για έναν αυτόματο μηχανισμό. Το λέω αυτό γιατί και στο Στρασβούργο αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση κρίσης και υπάρχει και το θέμα ιδιαίτερα του overbooking, όπου μετά γίνεται κλήρωση για το ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Θα πρέπει να ξέρουν οι επιβάτες πώς θα αποζημιωθούν μία τέτοια στιγμή. Να το ξέρουν εκ των προτέρων όμως, όχι τι τους προτείνει η εταιρεία εκείνη τη στιγμή διαφορετικά γίνονται διακρίσεις και υπάρχει άνηση μεταχείριση από πλευράς ε, ε, αερομεταφορέν. Ε, σας όλοι. Διαδικαστικό. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κύριο Κράμερ γιατί μίλησε για ομάδες που θα ήθελα να ξαναδούν τα επίπεδα αποζημίωσης. Εμείς θα ψηφίσουμε την τροπολογία του Προέδρου δηλαδή την 157, που υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Δεν ξέρω εσείς σε ποια ομάδα αναφέρεστε, αλλά όχι στην ομάδα των σοσιαλιστών, αυτό είναι σίγουρο. Michael, yeah, you're talking about the fact... Αναφέρεστε στο, στο, τι ισχύει στους σιδηροδρόμους σε σχέση με τις αεροπορικές μεταφορές για τη μία ώρα για παράδειγμα κτλ. Να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση αυτή. Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία θέλω να θίξω. Το πρώτο έχει να κάνει με τη συμβαστική ΚΕΙ. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε ενδυναμώσει τη διατύπωση στο σημείο αυτό. Με τη δική μου τροπολογία 157 στην οποία ουσιαστικά ήθελα να εξασφαλίσω ότι οι επιβάτες και στις δύο περιπτώσεις που ταξιδεύουν προς μια χώρα ή από μια χώρα έχουν τις ίδιες, τα ίδια δικαιώματα. Τόσο αναχωρούντες όσο και αφικνούμενοι. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι και στις δύο περιπτώσεις ε, οι επιβάτες αυτοί μπορούν να βρεθούν ε, με τα ίδια προβλήματα. Πάρα πολλές φορές ε, πρέπει πολύ γρήγορα να επιβαστούν οι αποσκευές προκειμένου να φύγει το αεροπλάνο και τελικά πολύ συχνά βλέπουμε ότι όταν φτάνει το αεροπλάνο στον προορισμό του οι αποσκευές μένουν απλώς ένα πολύ μεγάλο καρότσι και περνάει πάρα πολλή ώρα μέχρι τελικά να δοθούν στους επιβάτες. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε επιβάτες ε, αφικνούμενους οι οποίοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους αναχωρούντες. Ε, τώρα, όσον αφορά την τροπολογία 15, τη δική μου τροπολογία 15, ο κύριος Σπέρκινς αναφέρθηκε σε αυτήν. Ξέρετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε την καλύτερη νομοθεσία του κόσμου, αλλά αν δεν έχουμε τα απαραίτητα όργανα επιβολής νομοθεσίας αυτής, τότε απλώς χάνουμε το χρόνο μας. Επομένως αυτό το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα ήθελα τα όργανα αυτά επιβολής να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να κάνουν πραγματικά τη δουλειά τους. Ένας κάτοικος από τη δική μου περιφερειακή τη δική μου περιφέρεια είχε πρόβλημα με την KLM, έστειλε μια επιστολή στην KLM και η KLM του, απάντησε ότι ήταν ε, μια κατάσταση νοτέρας βίας και δεν μπορούσε να κάνει κάτι το συγκεκριμένο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καλούνται τα όργανα επιβολής να κάνουν εδώ πέρα τη δουλειά τους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από την επιβάτη αυτό να βρει το δίκαιο του αναγκαστικά μόνο με μια αεροπορική εταιρεία που μπορεί να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο Κίθ λοιπόν αναφέρθηκε σε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα όργανα επιβολής να κάνουν πραγματικά τη δουλειά τους, να επιτελούν πραγματικά το έργο τους. Και θεωρώ ότι δεν κάνουν κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Και αυτό περιλαμβάνει και την δική μου υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Κυρία Γέγκε. Let me first of all... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδες εισηγητές. Τον συγχαίρω για την εξαιρετική έκθεση. Εμείς με ικανοποίηση ε, συνεργαστήκαμε με τον εισηγητή. Πιστεύω πως έχουμε τους ίδιους στόχους και βεβαίως ε, στην αναθεώρηση του 261 θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες για τους επιβάτες και να έχουμε ενιαία εφαρμογή ε, του κανονισμού. Θα ήθελα να πω πως η Κομισιόν ε, επί της αρχής μπορεί να υποστηρίξει όλες τις συμβαστικές προτάσεις και τις ε, 30 ε, πλην της ΚΑΠΑ αποζημίωση για την καθυστέρηση αποσκευών κατά αναλογία με τις ανάγκες του επιβάτη. Δυστυχώς αυτό δεν καλύπτει από τη συνθήκη του Μοντρεάλ, οπότε μας περιορίζει η νομοθεσία, αλλά θεωρούμε πως οι συμβαστικές τροπολογίες αποτελούν μια καλή βάση και αναμένουμε αύριο μια θετική ψηφοφορία. Επίσης, σας δώσαμε πληροφορίες για την εκστρατεία των δικαιωμάτων επιβατών και το τι κάνει η κυρία Κούνεβα και περισσότερες λεπτομέρειες για τις εφαρμογές ε, ξυπνά τηλέφωνα. Δεν θα σπαταλίσω όλο το χρόνο σας, καθώς συμφωνούμε με τον εισηγητή. Να προσθέσω πως αυτή τη στιγμή κάνω μια αξιολόγηση αντικτύπου για την αναθεώρηση του 261 και η δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε το Δεκέμβριο είναι ανοιχτή μέχρι τις 11 Μαρτίου και θεωρούμε πως η έκθεση του κυρίου Τέιλορ θα αποτελέσει μια καλή βάση και θα εξεταστεί προσεκτικά στην αξιολόγηση αντικτύπου βεβαίως και η αναθεώρηση του 261 θα γίνει εκ με, το πακέτο με την οδηγία των ε, ταξιδιωτικών πακέτων. Επίσης η Κομισιόν εξετάζει τον κανονισμό 1008-2008 ε, για τα αεροπορικά ταξίδια, για το κατά πόσον προσαρμόζονται συνθήκες της αγοράς. Επίσης, να σας ενημερώσω για τις κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, για την εφαρμογή του κανονισμού 1108 για άτομα με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα. Συζητάμε τους ενδιαφερομένους, πρέπει να εκδοθούν μέχρι την άνοιξη του 2012 για να έχουμε μια εφαρμογή μέχρι τους παραολυμπιακούς αγώνες στο Λονδίνο. Αναμένουμε λοιπόν αύριο μια θετική ψηφοφορία και ε, ευχαρίστως να συνεχίσουμε την... το έργο μας πάνω σε αυτό το σημαντικό ζήτημα για όλους μας. Ευχαριστούμε. Κύριε Τέιλορ. Um, thanks, Ευχαριστώ Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω όλους για τα πολύ καλά σας λόγια. Δύο-τρία πράγματα θέλω να πω πολύ γρήγορα. Συμβαστική H. Ήταν μια κάποια πρόκληση να πετύχω συμφωνία για την τροπολογία αυτή. Πρέπει να σας πω ότι σχετικά με την τροπολογία αυτή θα πρέπει, είπαμε μάλλον, ότι ενδεχομένως να πρέπει οι οικογένειες με παιδιά να, να θεωρηθούν ως πρόσωπα με περιορισμένη κινητικότητα, PRM, και είπαμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες. Είναι σαφές στην έκθεση ότι θέλουμε μια βελτιωμένη πρόσβαση στις πληροφορίες και λέμε επίσης ότι υπάρχει στο σελίδα οι εκστρατείες που γίνονται σε ορισμένα κράτη-μέλη, καθώς επίσης και για αυτή την εφαρμογή για τα ΕΦΗ e κινητά τηλέφωνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έχουμε βέβαια και τα όργανα επιβολής και τις ίδιες αεροπορικές εταιρείες. Όλοι αυτοί οι φορείς θα πρέπει να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες και την κατάλληλη υποστήριξη. Εν τέλει λοιπόν πιστεύω ότι αν έχουμε επιβάτες αποκλεισμένους λόγω του χιονιού στο Έσεξ ή στην Εστονία σε κάποιο αεροδρόμιο θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπιστεί η κατάστασή τους πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν τα άτομα με αναπηρίε να μπουν στο αεροπλάνο με τον εξοπλισμό τους, για παράδειγμα με έναν σκύλο, αν ο επιβάτης είναι τυφλός. Πιστεύω επίση ότι ε, αν ε, τα όργανα επιβολή αντιμετωπίσουν πιο γρήγορα τι καταγγελίε των επιβατών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εγκρίνει τελικά τη συστάση έκθεση αυτή, τότε θα στεφθεί με επιτυχία το όλο εγχείρημά μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Και όπως ξέρετε τα θαύματα αργούν να γίνουν πραγματικότητα, αλλά μπορεί να γίνει και το θαύμα. Αύριο θα ψηφίσουμε και προβλέπεται συζήτηση στην Ολομέλεια του Μαρτίου για την αυριανή ψηφοφορία. Παρακαλώ πολύ μην ξεχάσετε να φέρετε τις κάρτε ψηφοφορίες. Το επόμενο σημείο στην μερίσια διάταξη είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Ο κύριος Κουμουτσάκος είναι συνσηγητής και ο κύριο Έρτουκ. Εισαγωγικά, όσον αφορά αυτή την πρώτη ενταλλαγή απόψεων, θα ήθελα να επενθυμίσω στου συναδέλφου ότι δύο συνεισηγητέ, θα συντάξουν μία ενιαία έκθεση, δεν θα καταλήξουμε με δύο διαφορετικές εκθέσεις. Μία έκθεση θα έχουμε. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στον κύριο Κομουτσάκο και στη συνέχεια στον κύριο Έρτουκα. Ο κύριος Κομουτσάκος λοιπόν έχει πρώτος το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια στιγμή λέει, κύριε Κομιτσάκο. Any subsequent meetings to the last discussion can be held outside. Αν θέλετε να συζητήσετε μπορείτε να περάσετε έξω για να ακούσουμε τον εισηγητή μας. Κύριε Κομιτσάκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως αναφέρατε, σήμερα έχουμε την πρώτη επίσημη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα όπως προτάθηκε από την Κομισιόν τον Οκτώβριο. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ το έργο μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω θέτοντας τα δίκτυα αυτά στην ευρύτερη στο ευρύτερο πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω της άνευ προηγουμένου κρίσης. Οπότε χρειαζόμαστε επιγόντω καλά νέα τα οποία θα στείλουν ένα θετικό μήνυμα το ότι δηλαδή η Ευρώπη μπορεί να κερδίσει το στοίχημα για αηφόρο ανάπτυξη. Η κρίση θα πρέπει να θεωρηθεί κίνητρο επενδύσεων και όχι εμπόδιο. Οι επενδύσεις στις ε, υποδομές των μεταφορών μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την κρίση και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Τα δίκτυα, οι ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, μπορούν να αποτελέσουν ένα εφαλτήριο για την αηφόρο ανάπτυξη που εκτιμούμε. Οπότε, έτσι, τα δίκτυα αυτά δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και πολιτική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά για το Κοινοβούλιο θεωρώ πως το 2012 πρέπει να αποτελέσει το έτος των διευρωπαϊκών δικτύων και είμαι πεπισμένος πως εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να γίνουμε η ατομομηχανή που θα επιτύχει αυτό το στόχο. Τώρα, για τη μέθοδο εργασίας, όπως είπε ήδη ο πρόεδρος, η έκθεση αυτή θα συνταχθεί και θα παρουσιαστεί από δύο συνεισηγητές, τον κύριο Ρτούγ και εμένα. Μία έκθεση λοιπόν θα υποβληθεί. Οπότε θα έχουμε τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις και βεβαίως ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν και τους ενδιαφερομένους στο μέτρο του δυνατού. Και βεβαίως θα ενημερώνουμε τους κοιόδες συγητές, την κυρία Μπαραντίγα, την κυρία Κράμερ, ε, Ζήλε και τον κύριο Κόλιτσεκ ενήμερους και θα συνεργαστούμε μαζί τους, οπότε θα οργανώσουμε συναντήσεις αργότερα. Επίσης θα συνεργαστούμε στενά με εισηγητές από τις Επιτροπές Αρμούδης... δηλαδή Περιβάλλοντος Περιφερειών και Εσωτερικής Αγοράς και εξυπακούεται, κύριε Πρόεδρε, πως θα συνεργαστούμε πολύ στενά με τους εισηγητές για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Στον αφορά τα επόμενα βήματα, μια ακρόαση για τις κατευθυντήριες γραμμές ε, που θα καλύπτει τρία σημαντικά ζητήματα, μεθοδολογία, διάδρομη και απαιτήσει έχει προγραμματιστεί για τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 8 Μαΐου. Ελπίζω να το εγκρίνουν οι συντονιστές. Και ελπίζουμε ο Επίτροπος ο κύριος Κάλλας να έρθει σε αυτή την ακρόαση. όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Η προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης ε, έχει προβλεφθεί για το τέλος Μαΐου. Μετά θα την παρουσιάσουμε τον Ιούνιο. Θα ψηφίσουμε το φθινόπωρο στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια μέχρι το τέλος του έτους ή αρχές του επόμενου. Όσον αφορά τώρα την ουσία του κανονισμού. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει ακόμα κανένα διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, μόνο διάφορα εθνικά. Λείπουν λοιπόν, ε, διάφοροι συνοριακοί σύνδεσμοι, υπάρχουν στενοποί στα σύνορα και οι κατευθυντήριες γραμμές μέχρι στιγμής είναι μόνο εθνικά ευχολόγια. Οι κυβερνήσεις σκέφτονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά η Ένωση και ειδικά το Κοινοβούλιο πρέπει να σκέφτεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, βάσει αυτά, εμείς, εγώ και ο κύριος Σερτούγ δηλαδή, καλωσορίζουμε την πρόταση της Κομισιόν ως μια καλή βάση για περαιτέρω εργασία. Βεβαίως, περιθώρια για βελτίωση υπάρχει για να εκαταστεί το έργο αυτό πιο φιλόδοξο και πιο ρεαλιστικό εκεί που πρέπει. Η πρόταση της ε, Κομισιόν, όπως είπα, είναι μια πολλά υποσχόμενη βάση για το περιττέρω έργο μας. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες ελλείψεις. Ως εισηγητές, σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με την άποψη και την προσέγγιση της Κομισιόν σε τομείς κλειδιά, ειδικά την προσέγγιση δύο ε, στρωμάτων με ένα συμπληρωματικό και ένα κύριο δίκτυο που θα βασίζεται βεβαίω και στις προτεραιότητες Ένωσης και των κρατών Συμφωνούμε επίσης με τις ε, απόψεις για μια σαφή προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί στις στενοπούς, στις διασυνοριακές διασυνδέσεις και την ε, διασύνδεση διαφορετικών μέσων μεταφορά και την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Πρέπει να υπάρξει καλύτερη διασύνδεση αεροδρομίων και σιδηροδρόμων και βεβαίω θαλασσίων ε, μεταφορών και λιμανιών ως ε, πύλαων προς τρίτες χώρες. Εδώ πέρα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στις λεωφόρους της θάλασσας ως σημαντικό συστατικό στοιχείο του δικτύου αυτού. Συμφωνούμε με τις απόψεις για καλύτερο συντονισμό και συνοχή των διαφόρων μέτρων και των μέσων χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των ευρωπαϊκών συντονιστών, των ευρωπαίων συντονιστών, είναι κέριος, αν και χρειάζεται βεβαίω κάποια διευκρίνηση. Η προτινόμενη προσέγγιση των διαδρόμων ως ένα μέσο διαχείρισης έχει επί της αρχής την στήριξή μας, αλλά θεωρούμε πως οι διάδρομοι αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν περισσότερο στο πλαίσιο των ε, κατευθυντηρίων γραμμών και όχι στο πλαίσιο του ΣΕΦ όπως έχει αυτή τη στιγμή. Επίσης, σαφής ε, και αυστηρότερη ερεσιμότητα, πράγματι επί της αρχής συμφωνούμε και συμφωνούμε με την αρχή ή το χρησιμοποιείς ή το χάνεις. Όσον αφορά τώρα τις ε, προθεσμίες, ε, έχουμε δύο προθεσμίες που προβλέπονται στον κανονισμό, 2030 για το βασικό δικτύο και 2050 για το συμπληρωματικό. Συμφωνούμε με αυτή την άποψη, αν και ξέρουμε πως τα κράτη-μέλη, οι συνάδελφοι, θα προτιμούσαν περισσότερη ευελιξία. Όσον αφορά το μέσο, δηλαδή τον κανονισμό. Εμείς ε, προτιμούμε την προσέγγιση της Κομισιόν, υποστηρίζουμε δηλαδή έναν κανονισμό αντί για κάτι το ασθενέστερο. Υποστηρίζουμε λοιπόν τον κανονισμό. Συνοψίζοντας η γενική μας ε, προσέγγιση είναι θετική όσον αφορά την πρόταση της Κομισιόν και βεβαίως κάποιες ρυθμίσεις και τροπολογίες οπωσδήποτε χρειάζονται. Και δεν έχω ψευδεστήσεις για το ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε πολλές διαφορετικές θέσεις και προτάσεις και βεβαίως θα είναι αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλοι. Αλλά για τα ακαθόδη ζητήματα, νομίζω ο καλός μου φίλος ο κύριος Ερτούγ ε, θα σας ενημερώσει. Εγώ κράτησα τα εύκολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. very much, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Κουμουτσάκο. Κύριο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Κουμουτσάκο. Ε, και για τα δύσκολα σημεία βεβαίως αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από την πρώτη εδώ πέρα, η οποία νομίζω είναι πάρα πολλά υποσχόμενη. Ε, έχουμε λοιπόν μια γενική ε, άποψη για το πώς ε, επιθυμούμε να είναι η ευρωπαϊκή πολιτική κινητικότητα. Ξέρετε, 2000 με 2008 αυξήθηκε κατά 8% η κινητικότητα και αυτό έχει οικολογικά και οικονομικά και κοινωνικά κόστη. Θα πρέπει λοιπόν στον τομέα των μεταφορών να έχουμε μία μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, καθώς μιλάμε για ένα 25% των εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μία ε, κοινωνία η οποία και ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου και τέλος βλέπουμε πως η ιστορική αγορά ολοκληρώνεται κάποια πράγματα πριν μπω τώρα στην ουσία, κάποιους αριθμούς ακόμα. Έχουμε 4,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα οδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2,5 ε, εκατομμύρια χιλιόμετρα ε, σιδηροδρόμων ε, και πολύ μικρότερο δίκτυο πλεύσιμων ποταμών. Γιατί το λέω αυτό, γιατί θα πρέπει να οδηγηθούμε πραγματικά σε ένα διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και θα συνδέονται όλες οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε κάτι που αφορά τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να γίνουν πιο ευρωπαϊκά στις σκέψεις τους και λιγότερο εθνικά θα ήθελα να αναφέρω τώρα σύντομα αυτό το οποίο ανέφερε και ο κύριος Κουμουτσάκος, το οποίο στηρίζω και εγώ. Πρώτα απ' όλα την προσέγγιση αυτή των δύο επιπέδων του βασικού και του πιο εκτεταμένου δικτύου. Αυτό θέλουμε πράγματι και εμείς και εμείς επίσης θεωρούμε πως θα πρέπει να έχουμε μια ρύθμιση με κανονισμό και όχι με οδηγία για να είναι πραγματικά δεσμευτικό το ότι θα γίνει. Επίσης η αρχή του είτε το χρησιμοποιήσει το χάνεις <laughs> και Έχουμε βεβαίως ε, και τη μεθοδολογία την οποία προτείνει η Κομισιόν. Τη μεθοδολογία, ναι, την υποστηρίζουμε συνάδελφοι, αλλά θα πρέπει να είναι αντικειμενική και αντιληπτή από όλους. Και βεβαίως ε, θα επανέλθω να σας πω πώς το βλέπουμε εμείς αυτό. Τέλος, υποστηρίζουμε, η ομάδα μου δηλαδή, την προσέγγιση της Κομισιόν πως θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο ότι θα πρέπει να είναι στο προσκήνιο η μετακίνηση με διαφορετικά μέσα, να καταργηθούν ή στενοποί και να έχουμε περισσότερες διασυνδέσεις και βεβαίως ε, όσον αφορά τις διασυνοριακές συνδέσεις που θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερες στο μέλλον από ό,τι σήμερα. Ο συνάδελφος ο κύριος Κουμουτσάκος σωστά ανέφερε το ποιες συζητήσεις θα έχουμε πιθανώς τους επόμενους μήνες, εβδομάδε και μήνες. Θα ήθελα και εγώ να το αναφέρω. Αναφέρθηκα στη μεθοδολογία. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό και το διαπιστώσαμε και στην συζήτηση μέχρι τώρα πως απαιτείται περισσότερη διαφάνεια και πληροφορίες. Αυτό ισχύει όχι μόνο για εμάς και όλους τους συναδέλφους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για τα εθνικά κοινοβούλια. Οι συνάδελφοι στα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα και να ψηφίσουν από αυτών των θεμάτων, οπότε χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Πρέπει επίσης να δούμε τη συζήτηση του τι θα γίνει με τις απαιτήσει σε υποδομές. Αναφέρονται στο έγγραφο αυτό το πώς θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις τεχνολογικές και λοιπές απαιτήσει. Και αυτό είναι σημαντικό για ολόκληρη την νομοθεσία. Κάτι άλλο επίσης σημαντικό, το οποίο βεβαίω και εγώ και ο συνάδελφος προσέξαμε και πρέπει να συζητήσουμε, είναι πως στο κύριο δίκτυο αυτή τη στιγμή δεν περιέχονται οι διάδρομοι εμπορευματικής μεταφοράς αγαθών είχαμε κάνει πριν από δύο χρόνια μία έκθεση. Νομίζω και αυτή οι διάδρομοι μεταφοράς αγαθών θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο βασικό δίκτυο. Ένα άλλο σημαντικό θέμα θα είναι το ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ποια είναι τελικά η δουλειά των συντονιστών και πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι πλατφόρμες των διαδρόμων και πώς θα λειτουργήσουν. Εδώ πέρα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, ειδικά με τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί και από τη σκοπιά τους βεβαίως έχουν τις ανησυχίες της επικουρικότητας για το ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο μπαίνει πάρα πολύ στα χωράφια των εθνικών αρμοδιοτήτων και θα πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να εξηγήσουμε με διαφανή τρόπο τα πράγματα για να ξεκαθαρίσουν αυτές οι παρεξηγήσεις που υπήρξαν. Επίσης πρέπει να συζητήσουμε το τι θα κάνουμε με τα διάφορα νέα έργα, τα οποία βεβαίως θα προκύψουν από τις διάφορες περιοχές, περιφέρειες, που βεβαίως περιέχουν και την μεθοδολογία που πρότεινε η Κομισιόν για το τι θέλουμε να κάνουμε με αυτά τα έργα και αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα το αντιμετωπίσουμε και τέλος ένα από τα σημαντικότερα ίσως το σημαντικότερο ζήτημα είναι η χρηματοδότηση συνάδελφοι Έχουμε τώρα την ιδιαίτερη κατάσταση ότι θα συνεργαστούμε και με τους ε, εισηγητές του μέσου συνδέοντας ε, την Ευρώπη και βεβαίως εκεί πέρα υπάρχει και η πρόταση της Κομισιόν η οποία προβλέπει 31,7 δισεκατομμύρια ευρώ και 10 ε, δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής και βεβαίως αντιλαμβάνομαι πως οι συνάδελφοί μας των λεγόμενων κλασικών χωρών της συνοχής έχουν εδώ πέρα τις επιφυλάξεις τους και αυτές τις επιφυλάξεις πρέπει να δούμε. Και εδώ πέρα πρέπει βεβαίως να είμαστε σε στενή συνεννόηση και με τις άλλες επιτροπές για να έχουμε μια κοινή και ισχυρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ε, μπορέσουμε αν χρειαστεί να αντισταθούμε και στο Συμβούλιο. Οπότε βεβαίω είμαι σίγουρο πω του επόμενου μήνε θα μα απασχολήσουν πολύ όλα αυτά και οι λεπτομέρειε. Ευχαριστούμε. Θα περάσουμε τώρα στου Κιώδη. Η κυρία Πιλμπάου πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι καταρχήν αποτιμούμε θετικά την πρόταση διότι το έγγραφο αυτό ορίζει τα προϋπάρχοντα προβλήματα τα οποία καταγράφαμε από τη δεκαετία του 80. Ε, όπως γνωρίζετε υπάρχει μεγάλη απόκληση ως προς τα διαθέσιμα στοιχεία μεταξύ κρατών μελών, μεγάλο κατακαιρματισμό και πολλά σημεία και πολλές στενοπούς. Γι' αυτό συμφωνούμε με την αναγνώριση των προβλημάτων και των στόχων που θέτει η Επιτροπή για να επιλύσει αυτά τα θέματα κατακαιρματισμού. Χρειάζεται λοιπόν επιγόντως να ορίσουμε μία σαφή και διαφανή στρατηγική, να ε, λάβουμε υπόψη και την διατροπικότητα. Επίσης θα πρέπει να ορίσουμε ένα ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να τηρούν και τα κράτη-μέλη γιατί, είναι, γιατί διαφορετικά θα είναι σαν να ξεκινούμε από το μηδέν. Επίσης να βελτιώσουμε την συνεργασία των κρατών μελών για ένα συντονισμό των σχεδίων για τα επενδυτικά σχέδια για να δούμε ποια είναι η τοπική και η περιφερειακή πραγματικότητα που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Θα πρέπει επίσης να έχουμε μία πρόβλεψη ρυθμιστικού χαρακτήρα. Να ορίσουμε προτεραιότητες όπως ορίζει το έγγραφο, αλλά παράλληλα θα πρέπει να καταβάλουμε μία προσπάθεια για να ορίσουμε τους δείκτες που χρησιμοποιούμε για τα κριτήρια αυτά, καθώς και ένα σύστημα μέτρησης αποτελεσμάτων. Όλα αυτά μας οδηγούν στην χρηματοδότηση. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με το δίκτυο Connecting Europe, με το μέσον αυτό. Θα πρέπει να ορίσουμε σαφείς στόχους, να προβούμε σε μια σαφή στοχοθέτηση, καθώς και κριτήρια επιλογής για να ορίσουμε αυτό το βασικό δίκτυο, δηλαδή ένα παγκόσμιο ε, δίκτυο και ένα διευρωπαϊκό. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό σύστημα και θα πρέπει να το προωθήσουμε. Τέλος, Θεωρώ ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται από τις επενδύσεις και από την επίλυση θεμάτων. Θα πρέπει να μας απασχολήσουν οι υποδομές μας, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να διακινδυνεύουμε, να αποτολμούμε παρά την κρίση. Έτσι, η πρόθεση των υποδομών θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να δράσουμε και στο παγκόσμιο δίκτυο. Δεν υπάρχουν απειλές μεταξύ κρατών μελών που έρχονται εκ των έξω και γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις υποδομές μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή το εξής. Ποιο ρόλο θα μπορούσαν να έχουν οι συντονιστές για την εκτέλεση και τον ρυθμό εκτέλεσης των προγραμμάτων, ποιες είναι οι απειλές και οι κίνδυνοι, έτσι ώστε τα κράτη να δεχτούν την πρόταση όπως ορίζεται. Δεν θα πρέπει να μας συμπιέζουν οι εθνικοί φόβοι, εθνικού καθαρά χαρακτήρα. Θα πρέπει να προωθήσουμε ευρωπαϊκά σχέδια τέτοιας εμβέλειας. <laughs> Uh, e, ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριο ζηλε Ζήλε. Κάθομαι εδώ πέρα άκρη-άκρη, αλλά με είδατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η θέση του ECR. Έχουμε κάποια εθνικά συμφέροντα τα οποία θέλουμε να εκφράσουμε. Θεωρούμε πάντως ότι υπάρχει μια συμβαστική πρόταση η οποία μπορεί να μας βρει σύμφωνος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει το κείμενο αυτό κανονισμός και να μην γίνει απόφαση στην περίπτωση αυτή που θα είναι κανονισμός δηλαδή θα είναι πολύ πιο δεσμευτικό το κείμενο αυτό και θα επηρεάσει ακόμα και τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τους σιδηροδρόμους στα πλαίσια της δημιουργίας των διαδρόμων. Είναι πολύ σημαντικός επίσης ο ρόλος των συντονιστών. Αν πραγματικά θέλουμε να πραγματοποιηθεί το σχέδιο αυτό με τους ε, διαδρόμους, θα πρέπει να αυξηθούν και οι ικανότητες των συντονιστών. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε μόνο για μια προσέγγιση σε δύο επίπεδα, αλλά σε τρία επίπεδα. Γιατί έχουμε το κεντρικό δίκτυο, το εκτεταμένο δίκτυο, αλλά και ένα δίκτυο που έχει να κάνει με τους ε, διαδρόμους που κατά την άποψή μου ουσιαστικά αποτελεί αυτό τη σωστή προσέγγιση. Κάτι που είναι σημαντικό για τα νέα κράτη-μέλη, ότι είναι κάτι το αμφιλεγόμενο, είναι η συμπερίληψη των ταμείων συνοχής στα πλαίσια της διευκόλυνσης του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη για τη χρηματοδότηση των διαδρόμων. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο όμως μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα στις χώρες που αποφελούνται από τα Ταμεία Συνοχής. Διαφορετικά στις χώρες αυτές δεν θα δούμε καθόλου νέα έργα και προγράμματα στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Κάποιες πολύ σημαντικές βέβαια ανησυχίε είχα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και από την πλευρά του Συμβουλίου. Στις σχετικές ομάδες εργασίας βλέπουμε ότι υπάρχουν πλέον κάποιες εξελίξεις κάποιες απόπειρες γίνονται προκειμένου να καταρριφθεί η ιδέα αυτή των διαδρόμων. Μιλάνε κυρίως για core network projects, για κάποια έργα, προγράμματα του κεντρικού, του βασικού δικτύου. Αυτό λοιπόν προκάλεσε ανησυχία, ιδίως ε, για τη δική μου την περιοχή, για τις βαλτικές ε, χώρες. Θα παρακολουθήσουμε πάντως εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση. Γίνονται λοιπόν κάποιες απόπειρε, όχι μόνο για να εξαλειφθούν τα, οι διάδρομοι και να έχουμε απλώ κάποια έργα, αλλά προβλέπεται και μία επέκταση του κεντρικού δικτύου σε, κάποια, σε κάποιους άλλους διαδρόμους με μία διαφορετική γεωγραφική κατανομή. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τις ε, βασικές ιδέες που εκφράζονται στο άρθρο 7 και δεν θα καταφέρουμε τελικά να έχουμε μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στο όλο εγχείρημα. Θα εξυπηρετηθούν μόνο τα συμφέροντα ορισμένων ε, χωρών, τρίτων κρατών. Και στο υφιστάμενο σχέδιο δεν καλύπτονται ορισμένες χώρες όπως για παράδειγμα η Ρωσία. Θα μπορούσαμε τέλος πάντων να βρούμε μια συμβαστική λύση, θα θέλαμε όμως η συμβαστική αυτή πρόταση να μην πάρει την μορφή που είχαμε δει, όπως για παράδειγμα τον Ιανουάριο με τους σιδηροδρόμους με την πρόθεση εκείνη που ακουστεί για τους σιδηροδρόμους με τη Ρωσία. Πολύ συχνά στις βαλτικές χώρες βλέπουμε ότι υπάρχει μία παραμέληση όσον αφορά το ζήτημα των σιδηροδρόμων. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες μεγάλες σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στην Ανατολική και την Δυτική Ευρώπη που φτάνουν για παράδειγμα γραμμές αυτές μέχρι τη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, αλλά πρέπει να συντοπίσουμε ότι σαφώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε και την Ρωσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε κάποιες βασικές ιδέες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μιλάμε για τα χρήματα των Ευρωπαίων ε, φορολογούμενο, με συγχωρείτε, και θα πρέπει να καταφέρουμε να επενδύσουμε τα χρήματα αυτά σε έργα τα οποία θα ωφελήσουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πιο ισχυρή όσον αφορά την πολιτική μεταφορών. Α μην ξεχνάμε λοιπόν και αυτή τη διάσταση. Ευχαριστώ. Sorry, Michael, να σα είχα πρώτα το λόγο σε εσά. Η πρόταση της ε, Κομισιόν είναι έξοχη στην περιγραφή του προβλήματος, αλλά πολύ κακή στην ανάλυση. Και όταν δουλεύει κανείς 20 χρόνια στα διευρωπαϊκά δίκτυα και δεν έχει επιτύχει τίποτα, τι έχουμε. Διάφορα μπαλώματα και πού είναι το κενό στα σύνορα. Έχει αποτύχει ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτή η ανάλυση δεν υπάρχει. Ναι εντάξει δεν υπάρχουν λεφτά. Αλλά είναι ίσως λανθασμένο το ότι σκεφτόμαστε τις μεγάλες γραμμές ε, Παρίσι, Μπρατσλάβα. Γιατί τι σκέφτονται τα κράτη-μέλη, ε, υπάρχουν ένα-δύο δισεκατομμύρια, τα παίρνουμε. Αλλά Βερολίνο, Νιρεμβέργη παραδείγματο χάρη, θα γίνει μόνο εάν υπάρχει γερμανική χρηματοδότηση. Το ίδιο και άλλα ενδογερμανικά ε, δρομολόγια, αλλά διασυνοριακά π.χ. Φράιμπουργκ και Κολμάρ, ανατείναξαν οι Γερμανοί υποχωρώντας τη σιδηροδρομική γέφυρα. Δηλαδή, πόσα χρόνια έχουν περάσει από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν έχει ξαναχτιστεί η γέφυρα. Βερολίνο και Φρότσλαβ. Το ίδιο. Ε, ήτανε, χρειαζόταν 2,5 ώρες στο Μεσοπόλεμο, σήμερα χρειάζονται 6 ώρες. Που έχει μεσολαβήσει και ο εξηλεκτρισμός της γραμμής. Και λένε, πως δεν χρειάζονται ε, λεφτά. Και σκεφτόμαστε διάφορα εκεί πέρα να γεφυρώσουμε το στενό της Μεσίνας και διάφορα τέτοια πράγματα. Και αυτό δεν αλλάζει και σε αυτήν εδώ πέρα την πρόταση. Πρέπει να αναλύσουμε καλύτερα. Οπότε έχουμε αφενός τον στόχο 20-20. Αναφέρθηκε ήδη πως ε, οι μεταφορές ε, συνεισφέρουν 30% ε, στις ε, εκπομπές. Τι γίνεται δηλαδή, ε, από τη μία μειώνονται οι εκπομπές της βιομηχανίας και από την άλλη ό,τι μειώνεται το ακυρώνουν οι μεταφορές. Να σας δώσω ένα νούμερο από τη Γερμανία. Το 1994 από όταν μεταρρυθμίστηκαν οι σιδηρόδρομοι έχουν πάει 40 δισεκατομμύρια στις μεγάλες αποστάσεις. Το αποτέλεσμα σήμερα 20% λιγότερο επιβάτες. Το αποπέδι δε οι, κοντινές ε, αποστάσεις έχουν αυξηθεί κατά 5% οι επιβάτες. Είμαστε τρελοί να ρίχνουμε τα λεφτά εκεί που δεν ταξιδεύει ο κόσμος και εκεί πέρα όπου υπάρχει η μεγάλη επιτυχία ε, η μεγάλη επιτυχία. επίση 90% των ε, σιδηροδρομικών μεταφορών είναι τοπικέ μεταφορέ κάτω από τα 50 χιλιόμετρα. Αυτή λοιπόν πρέπει να είναι η προτεραιότητα και δεν υπάρχει εδώ πέρα. Εάν λοιπόν ξεκινάμε από το ότι ναι βεβαίως ε, δεν υπάρχει εθνικό ενδιαφέρον για δύο συνοριακές μεταφορές τότε πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο και να δώσουμε ακριβώς προτεραιότητα στα κομμάτια εκείνα τα διασυνοριακά. Και να μην πάμε από ένα 20% στο 30%, αλλά να πούμε πως εκεί πέρα βρίσκεται η προσθέμενη αξία. Τα 37 χιλιόμετρα στις δύο πλευρές των ε, σύνορων να τα χρηματοδοτήσουμε μέχρι 60% να τα συγχρηματοδοτήσουμε. Έτσι θα έχουμε μεγαλύτερο ευρωπαϊκό αποτέλεσμα. Αν συνεχίσουμε όπως τώρα θα πάρουν τα λεφτά τα κράτη-μέλη για αυτά τα οποία τους ενδιαφέρουν, δηλαδή τα εθνικά δρομολόγια και η Ευρώπη δεν θα παίξει κανένα ρόλο. Τώρα για τα υπόλοιπα τα διευρωπαϊκά δίκτυα και μεγάλες ε, μεγάλες διαδρομές και θόρυβο κτλ. Κοιτάξτε, εάν δεν θέσουμε τις σωστές ε, προτεραιότητες πάλι θα αποτύχουμε και μετά από λίγα χρόνια δεν θα έχει συμβεί πάλι τίποτα και αυτό θα είναι πραγματικά κρίμα. Ευχαριστώ. Κύριε Σκόλτσεκ. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ ορισμένα σχόλια. Ο συνάδελφος από τις βαλτικές χώρες βλέπει τη διάσχεση τη διάσταση βορρά-νότου. Όμως για την ε, τσεχική δημοκρατία υπάρχει και η ε, διάσταση ε, Ανατολής και Δύσης. Δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτό που είπε ο συνάδελφος. Οι Γερμανοί θέλουν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας, ας πούμε, από τη Δρέσδη. Και δεν τους ενδιαφέρει η τσεχική επικράτεια, κοιτά να την παρακάμψουν. Άρα η διατροπικότητα δεν λαμβάνεται υπόψη παρκώς. Στις χώρες ε, Μπενελούξ έχουμε τη Γαλλία ε, από ε, προς το βορρά. Αλλά αν δούμε προς Ανατολά στη Βιέννη και την περιοχή του Δούναβη, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες μεταφορές και ούτε και προβλέπονται. Δεν μας ενδιαφέρει η χρήση του Δούναβη στα πλαίσια των εσωτερικών μεταφορών, των ποτάμιων μεταφορών. Έχουμε δύο διόδους από το Βερολίνο προς Ανατολάς, η άλλη προβλέπεται από το Μόναχο και τελειώνει στη Βουδαπέστη και στο ενδιάμεσο υπάρχει μαύρη τρύπα, δηλαδή η τσεχική δημοκρατία. Εάν λάβουμε υπόψη αυτό το κριτήριο σοβαρά, δηλαδή την σύνδεση των ε, ε, πρωτευουσών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις, όλους τις ε, διάβλους για να, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε την Ευρώπη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις υποδομές, να μιλήσουμε και για τα σχέδια TEN. Η περιφερειακή συνεργασία είναι ύψης της σημασίας ιδιαίτερα ε, για ε, τις ε, υποδομές που δεν περιλαμβάνονται στο TEN-T. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και περιφερειακούς διαδρόμους μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, διασυνδεσιμότητας. Έτσι θα δούμε αν υπάρχει πραγματικά ή όχι. Έχω 14 ομιλητές στον κατάλογο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι θα γίνουν και άλλες συζητήσεις επί του θέματος και μία ακρόαση. Δύο λεπτά λοιπόν ο καθένας και σας παρακαλώ να είσαστε πειθαρχημένοι κατανοώ ότι στο Κοινοβούλιο, ε, αν και όλα έχουν προϋποθεί, δεν έχουν προϋποθεί από όλους. Αλλά θα ήθελα να αντισταθείτε σε αυτό τον πειρασμό. Δύο λεπτά έκαστος. Αρχίζοντας από τον κύριο Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι πολύπλοκο, η στιγμή είναι δύσκολη και συνολικά οι εμπειρίες του παρελθόντος δεν είναι ε, τόσο απεσιόδοξες όπως τις περίγραψε ο κ. Κάμερα, αλλά ούτε τόσο θετικές. Μπορούμε να το δούμε και διαφορετικά. Εγώ δεν θα ήμουν τόσο αρνητικός. Υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα. Το ένα λέει να πάρουμε τα λεφτά από τα διευρωπαϊκά δικτύα και να πούμε στο και να πούμε πως οι μεταφορές δεν τα χρειάζονται αυτά τα λεφτά. Νομίζω πως ε, τα λάθη του παρελθόντος θα πρέπει να τα δούμε και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Πρώτον, πρέπει να κάνουμε κάτι με το ΣΕΦ. Δεύτερον, θα πρέπει να ε, αφήσουμε τα νούμερα και να έχουμε περιορισμένους συγκεκριμένους στόχους. Αλλά θα πρέπει νομίζω να μπορέσουμε να πάμε και στο Συμβούλιο Μεταφορών και να πούμε πως υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή συνοχή η οποία είναι για μας ένα σημαντικό στόχος. Επίσης θα πρέπει να δούμε τις επενδύσεις των μεταφο στις μεταφορές ε, ως κάτι το οποίο είναι διπλά καλό. Πρέπει να το πούμε και στους συναδέλφους στην Οικονομική Επιτροπή πως αυτά δεν είναι λεφτά τα οποία αφαιρούμε από άλλους αλλά είναι λεφτά τα οποία οδηγούν σε μια πιο αηφόρο οικονομία, σε μια πιο αηφόρο κινητικότητα και δεύτερον πως μπορούν να εξυπηρετήσουν όλες τις περιφέρειες και βεβαίως αν έχουμε και την αρχή ε, της ε, επικουρικότητας αλλά και της ερεσιμότητας Νομίζω πως θα μπορέσουμε να αποφύγουμε πάρα πολλά λάθη του παρελθόντος, το δηλαδή δίναμε λεφτά χωρίς να εξετάζουμε το τι γινόταν και το εάν υπήρχε κάποια ευρωπαϊκή προστομήνη αξία. Οπότε η πρότασή μου, κύριε Πρόεδρε, ε, από πλευρά και της ομάδας μας, είναι να έχουμε συγκεκριμένα θέματα, να είμαστε ε, επικεντρωμένοι και βεβαίως αυτό το οποίο μας προσφέρει η Κομισιόν και είναι πάρα πολύ θετικό να το εκμεταλλευτούμε. Γνωρίζουμε το παρελθόν, γνωρίζουμε τα λάθη που γίνουμε. Νομίζω πως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις εδώ πέρα χωρίς να α, μπω σε πολλές λεπτομέρειες γιατί ξέρω πως δεν θα είναι αυτή η τελευταία μας συζήτηση αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνεπτικοί. Κύριε Αλχαντραουή, μπορείτε να περιοριστείτε κι εσείς. Θα προσπαθήσω. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως πρέπει να απομακρυνθούμε από το σκεπτικό που είχαμε μέχρι σήμερα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Πράγματι, η επένδυση σε αυτά τα δίκτυα αποδίδει αμέσως και εμέσως και μπορεί να αποτελέσει έτσι και μια διέξοδο για την ε, κρίση και βεβαίως θα πρέπει να δούμε πως θα έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Η μεθοδολογία αναφέρθηκε, νομίζω πως είναι ένα πρώτο βήμα όπου ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε σαφήνεια εμείς ως ε, κοινοβούλια και θα πρέπει πράγματι να οργανωθούμε για να υπάρξει μια σωστή αντίληψη και να αποφύγουμε και τις πολλές ε, τροπολογίες αργότερα Οπότε νομίζω πως είναι πάρα πολύ καλή, εξαιρετική ιδέα να οργανωθεί μια κρόαση. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε το ότι θα έχουμε μια σκληρή αντιπαράθεση με τα κράτη-μέλη όσον αφορά ακριβώς τους όρους που θέτουμε για την ε, χρηματοδότηση. Δυστυχώς θα πρέπει να μπορέσουμε να ελιχθούμε και να περιοριστούμε πράγματι στα έργα εκείνα τα οποία θα έχουν ευρωπαϊκή προσθέμενη Να δούμε λοιπόν τι θα χρηματοδοτήσουμε με ποιε προθεσμίε, αλλά να υπάρχει και μια τεχνολογική διαλειτουργικότητα. Δεν έχει κανένα νόημα να ρίχνουμε ευρωπαϊκά λεφτά σε κάτι το οποίο δεν λειτουργεί διεθνώ και διασυνοριακώ. Θα συμφωνήσω δε με του συναδέλφου που είπαν πω ε, πρέπει να πείσουμε και τα εθνικά κοινοβούλια να δούμε πώς θα γίνει αυτός ο διάλογος ε, για να είναι μαζί μας και τα Εθνικά Κοινοβούλια και τέλος η μεγάλη σημασία της ε, άλλης έκθεσης για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη και το πακέτο μέσων που θα έχουμε για να μπορέσουμε να επενδύσουμε γιατί βεβαίως χωρίς λεφτά δεν γίνεται τίποτα και πρέπει να αναπτύξουν μια στρατηγική και με την Επιτροπή μας και με το υπόλοιπο Κοινοβούλιο για να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε με, για το πώς θα μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε αυτά τα 31,7 δισεκατομμύρια ευρώ και με το ΣΕΦ και με τις κατευθυντήριες γραμμές. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Mr. Ο κύριος Ντεμπάκε, δύο λεπτά. Μπορείτε να περιοριστείτε δύο λεπτά. Τα κατάφεραν οι προηγούμενοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μας σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένη με την ε, πρόταση αυτή. Να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το Κοινοβουλίο μας θα πρέπει να δώσει ένα μήνυμα για το ότι διαλέγουμε μια ευρωπαϊκή πρόπτικη. Ξέρω πως θα έχουμε δύσκολη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά για το Κοινοβούλιο μας θα πρέπει και εμείς ως βουλευτές να έχουμε μια προοπτική ε, όσον αφορά την ε, άποψη την οποία θα παρουσιάσουμε. Και θεωρώ πως τα ε, υφιστάμενα δίκτυα μεταφορών δεν επαρκούν, βλάπτουν την οικονομία μας και θα πρέπει να υπάρξει μια συνεκτική πολιτική ανάλυση Βεβαίως ε, υπάρχει μια οικονομική ε, κρίση και θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τους συντάκτες της έκθεσης του μέσου συνδέοντας ε, την Ευρώπη και να δούμε το ότι θα γίνει όχι μόνο με τη δημόσια αλλά και την ιδιωτική χρηματοδότηση ως ένα είδος μόχλευσης, κάτι το οποίο έχει κρίσιμη σημασία για την μελλοντική ανάπτυξη. Και κάτι άλλο, ίσως κάπως ε, δευτερεύω, νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία με τους ε, συντονιστές. Αυτά και τελειώνω εδώ πέρα. Ευχαριστούμε. Λίχτενμπεργκερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κάποιες ε, παρατηρήσεις να προσθέσω και εγώ. Εξακολουθώ να βλέπω ένα μοιραίο κόλλημα με μεγάλα έργα, πολύ μακροπρόθεσμα και δημιουργούν προβλήματα σε καιρούς οικονομικής κρίσης όπου ακόμα και ένα σχετικά πλούσιο κράτος όπως η Αυστρία θα πρέπει να αναβάλει κάποια έργα γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για χώρες οι οποίες ε, έχουν πολύ ε, μεγαλύτερες δημοσιονομικές πιέσεις από την Αυστρία. Τώρα, αν δούμε όλα τα μέσα τα οποία θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να χρηματοδοτήσουμε πράγματα τα οποία εντάξει πολύ, πολύ ωραία να λειτουργήσουν ίσως μετά τον θάνατό μας, αλλά δεν θα υπάρχουν τα μικρά για τα οποία χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε Αυστρία και αλλού και στην Ελλάδα πως ε, μεταφέρουν αυτή τη στιγμή τα δίκτυα λιγότερα αγαθά και ανθρώπους γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για την λειτουργία τους τώρα. Οπότε θα πρέπει να δούμε να κάνουμε το εφικτό τώρα, αυτή τη στιγμή και να επιφέρουμε μικρότερες βελτιώσεις ε, στα υφιστάμενα ή να φτιάξουμε μικρότερα κομμάτια δικτύων που θα οδηγήσουν σε άμεσες όμως βελτιώσεις της υποδομής. Αυτό το κόλλημα στα μεγάλα έργα έχει και έναν άλλο κίνδυνο. Ένας ομιλητής το ανέφερε ήδη. Πως για να γίνει αυτό πρέπει να περιορίσουμε την ε, ελευθερότητα. Αν είχε πάει κανείς στη Βάλτε Σούζα και μιλούσε με τους ντόπιου και είδη το τι είχαν κάνει εκεί πέρα, αυτό ακριβώς αποδεικνύει αυτή την αρχή. Δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν ε, ανησυχίες για το περιβάλλον, ανησυχίες των ανθρώπων και τα παραμελούν όλα αυτά, γιατί θέμε όπως και δίποτε όχι να κάνουμε βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου, αλλά νέο μεγάλο έργο. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε ένα σημείο ακόμα. Βλέπω πως ε, τα διαφορετικά μέσα, η διατροπικότητα ε, είναι σημαντικά αλλά βλέπω πως δικαιολογούνται, ε, αποτελούν δικαιολογία για τη χρηματοδότηση αυτοκινητοδρόμων που δεν θα ε, χρηματοδοτούνταν τόσο εύκολα. δεν υποστηρίζω λοιπόν αυτή την τάση. Ευχαριστώ. Κύριος Φαντάλεν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι το θέμα αυτό είναι μεγάλο τεστ και για εμάς, για τα μέλη της Επιτροπής μας. Γιατί όλοι λένε για το πόσο σημαντική είναι η σύνδεση στη δικιά του χώρα. Αλλά μιλάμε πως ε, θα πρέπει να έχουμε ε, ένα βασικό δίκτυο και εδώ πέρα ακούμε το πώς θα συνδεθεί η κομμόπολη Φράιμπουργκ με το χωριουδάκι που λέγεται Κολμάρ. Ε όχι, να μιλάμε για πραγματικές συνδέσεις που έχουν κάποια σημασία για τους Ευρωπαίους και ένα σημαντικό αριθμό επιβατών. Εδώ πέρα λοιπόν είναι πραγματικά που θα κρυθεί η Επιτροπή μας και τα μέλη της. Τώρα, ε, για τους ε, λιμένες, τους ε, θαλάσσιους. Δεν ξέρω αν χρειάζεται πραγματικά για όλα αυτά τα λιμάνια να δώσουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και κάτι άλλο. Ε, μπορεί κάποιες ομάδες να μην είναι υπέρ των, ε, της εσωτερικής ε, ναυσιπλοείας. Εγώ χαίρομαι για το ότι επιτέλους έχει μεγαλύτερη προσοχή και αυτός ο κλάδος. Ευχαριστώ κύριε κύριο κύριος Κάντσιαν. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά για αυτό το θέμα και ελπίζω να έχω και άλλες ε, δυνατότητες να μιλήσω χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες. Θα το κάνω αργότερα. Νομίζω ότι η Επιτροπή έκανε, ε, επιτέλεσε ένα εξαιρετικό έργο χωρίς να λάβει υπόψη όλες τις επιθυμίες, αλλά προώθησε μία ε, αξιόπιστη εργασία γιατί όσον αφορά το Μπρένερο και τη σύνδεσή του θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί εκ των προτέρων. Δύο θέματα ως προς τη μεθοδολογία καταρχήν. Βλέπω ότι η Επιτροπή από τον Οκτώβριο του 2008 το είχε συζητήσει και είναι σαφής η έννοια του διαδρόμου, όπως ορίστηκε. Μιλάμε για ένα τρίτο επίπεδο προγραμματισμού. Πολλοί έτσι το θεωρούν, αλλά πρόκειται για ένα βασικό στοιχείο διακυβέρνησης. Νομίζω λοιπόν ότι και οι διάδρομοι αυτοί θα πρέπει να περάσουν από ρόλο διευκολυντών σε ε, ρόλο αρχών. Θα πρέπει να ορίσουμε τις ε, προτεραιότητες και μέσα στα πλαίσια των TNT για το εγγύς μέλλον. Ως προς το ΤΣΕΦ μιλάμε για το 2012-2020, το μέσο σύνδεσης για την Ευρώπη, ναι το Connecting Europe δηλαδή. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την, ε, την ε, χρήση των project bonds και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να εφαρμόσουμε ορισμένες αρχές άμεσα και να μην περιμένουμε την έγκριση του μέσου Connecting Europe. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την παρούσα κρίση και να αρχίσουμε τα σχέδια άμεσα, δηλαδή να προβούμε σε μια σαφή ιεράρχηση. Αντώνιο, θα γίνουν ε, πολύ περισσότερες συζητήσεις και θα γίνονται για τους επόμενους έξι μήνες. Λάχτφριντ, για δύο λεπτά. Προβλέπετε και ακρόαση, όπως ξέρετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω πράγματι να μην επαναλάβω αυτά τα οποία ε, ακούστηκαν ε, ήθελα να πω πως ε, στον κύριο Τσίλε δεν κάθεται άκρα αριστερά, κέντρο αριστερά, άκρα αριστερά. Ε, είμαστε Ε, τέλος πάντων είναι και μία πρόοδος ε, να σας βλέπουμε εκεί πέρα. Τώρα. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, να μου δώσετε το χρόνο μετά που έχασα από το θόρυβο. Λοιπόν, συγκεκριμένα τώρα για το θέμα μας. Το σημαντικότερο είναι ε, πως ε, συμφωνούμε με τον κύριο Κράμερ πως πρέπει να ε, υπάρχει ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Συμφωνούμε με τον κύριο Κράμερ. Εκεί που δεν συμφωνούμε είναι η σχέση που παρουσίασε μεταξύ τοπικών δρομολογίων και μεγάλων αποστάσεων θεωρώ πως ειδικά όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία οι μεγάλες αποστάσεις ε, γιατί εμείς λέμε πως πρέπει να φύγουν ακριβώς οι μεγάλες και βαριές εμπορευματικές μεταφορές από τους αυτοκινητόδρομους και να πάνε στους σιδηρόδρομους. Είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει αυτούς τους ε, διαδρόμους τους σιδηροδρομικούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά βεβαίω και για τις επιβατικέ μεταφορές για να αποτελέσουν ανταγωνισμό πραγματικές τις ε, πτήσεις και στους αυτοκινητοδρόμους και δεν είναι τόσο άσχημη η πρόταση της Κομισιόν, μπορούμε να τη δούμε στις λεπτομερίες τους, αλλά οι μεγάλοι αυτοί οι άξονες βορρά-νότου είναι νομίζω καλοί, είναι επίσης συνδέσεις διασυνοριακές και συμφωνούμε όλοι πως ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για εθνικά ε, έργα αλλά να φορούν περισσότερες χώρες και ακριβώς δεν έχει νόημα να εγκρίνουμε εμείς κάποιο διευρωπαϊκό δίκτυο και μετά να μην κάνουν τίποτα τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε και μετά στις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους από τους φιλελεύθερους. Σε ένα λεπτό, λοιπόν, να πω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ανακτήσει την οικονομική της ανάπτυξη και έχουμε ένα κίνδυνο απόκλησης ανάμεσα στο βορρά και στο νότο της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, η οποία θα πρέπει να διέπει τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε και επίσης να έχουμε και μια ανάλυση κόσμου ωφέλους για να επιλέξουμε τα σωστά έργα. Ευχαριστούμε πολύ. Ντουράν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Καταλαβαίνω απόλυτα την μέθοδο των δύο επιπέδων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που σχολίασαν οι δύο συνάδελφοι να επιστήσω την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάτι που θεωρώ ότι υπάρχει μια, υπάρχει μια ανομαλία όσον αφορά την, επίλεξη των, την επιλογή των πόλων για το κεντρικό δίκτυο. Δεν αναφέρομαι στις μικρές πόλεις, αλλά σε αυτές που πραγματικά μπορούν να, προσ, να προσθέσουν μια σημαντική προστιθέμενη αξία. Και αναφέρομαι για παράδειγμα στην Λιέγη. Πρόκειται για την πόλη που έχει ένα πολύ σημαντικό το τρίτο σε σειρά εσωτερικό λιμάνι με πάρα πολλές πάρα πολλά φορτία που φτάνουν. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κόμβο. Πρόκειται για ένα πολυτροπικό α, λιμάνι τη όλη περιφέρεια. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια ανομαλία στο σημείο αυτό. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό στο κεντρικό δίκτυο να έχουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο που πηγαίνει από την Άβρα στην Κολονία, περνώντα από τη Βαλονσιέν. Θεωρώ λοιπόν ότι τα δύο αυτά στοιχεία έχουν μια πραγματική προστιθέμενη αξία και θα πρέπει να ενταχθούν στο κεντρικό δίκτυο της πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ. Πέρκερ, παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω την ιδέα της Κομισιόν να υπάρχει μια προστιθέμενη αξία, δηλαδή να γίνει προσπάθεια μιας ευρωπαϊκής οργάνωσης και συντονισμού να έχουμε ένα συνολικό έργο όταν μιλάμε για αυτούς τους διαδρόμους. Ο διάδρομος Βαλτικής Αδριατικής είναι ένα καλό παράδειγμα να συνδεθεί η Βαλτική με την Αδριατική και να έχουμε μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Είναι μια προτεραιότητα που προβλέπεται. Αυτό το οποίο επίσης θεωρώ είναι πως από την αρχή και γι' αυτό παρακαλώ τους ε, συντάκτες να μπορέσουμε να παραμερίσουμε τα εμπόδια που έχουμε τώρα για να μπορεί να πάει κανείς ε, από το Ταλίν μέχρι την ε, Αδριατική με το τρένο. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα ηλεκτρικού ρεύματος, ασφαλείας κτλ. κτλ. Δεύτερον, γνωρίζουμε πως είναι δύσκολο να περάσουν τα έργα, τα μεγάλα έργα υποδομών αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει επιβαρύνσεις λόγω αυτών των δικτύων να κάνει και τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού, δηλαδή προστασίας από θόρυβο και να τα συγχρηματοδοτεί για να υπάρχει και αποδοχή από τον τοπικό πληθυσμό. Και το επόμενο πρέπει όπως ε, προβλέπει και η Κομισιόν να υπάρξει ένας Ευρωπαίος συντονιστής ο οποίος θα ε, φροντίζει τα λεφτά αυτά να πάνε όντως για τα έργα τα οποία προβλέπονται και να υπάρχει ακριβώς η διασυνοριακή αυτή διάσταση και ο έλεγχος ευθύς εξ αρχής γιατί Βεβαίω, ο έλεγχος είναι καλύτερος από το να βασιζόμαστε μόνο στην εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω το ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους εθνικούς εγωισμούς και τις διελκυστίνδες μεταξύ γειτόνων για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα και τις στενοπούς. Θα ήθελα να πω ότι από όσα άκουσα από τον εισηγητή θα ε, εισαγάγουμε τους διαδρόμους της guidelines σε σχέση με το μέσο Connecting Europe. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο θα ορίσουμε ξεχωριστούς κανονισμούς έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα σετ, σε μια σειρά χαρτογραφήσεων σε σχέση με τους διαδρόμους. Και δεν ξέρω κατά πόσο η Επιτροπή θέλει να προβεί σε αυτή την επακριβή χαρτογράφηση. Κύριε Κουμουτσάκο, μπαίνετε στη σε μια μεθολογία την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε βεβαίως, την έχουμε υποστηρίξει καταρχήν, όμως επισέρχονται στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Μιλάμε για το άρθρο 59, δηλαδή οι αποσύρσεις θα την χάνουν κυρώσεων, ναι ή όχι. Αυτό θα πρέπει να το ορίσουμε εκ νέου. Ως προς την αναθεώρηση Υπάρχει αρχή use it or lose it, όπως ορίζει η ενδιάμεση αναθεώρηση ή όχι. Τι γίνεται ως προς την ευελιξία προθεσμιών. Θα πρέπει να μας πείτε κύριε ε, Κουμουτσάκο τι εννοείται όταν μιλάτε για ευελιξία προθεσμιών. Και ως προς τους ε, διάβλους εμπορευμάτων, και τις εμπορευματομεταφορές θα πρέπει να ξέρουμε ε, ε, επακριβώς τι εννοούμε για να μην υπάρχει αποκλεισμός διαδρόμων. Τι θα γίνει με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις κύριε Κουμουτσάκο έναντι της Κομισιόν μπορούμε να επανέλθουμε ως προς ορισμένα σχέδια υποδομών. Θα ήθελα να ρωτήσω και την Επιτροπή τι γίνεται με τον εκτελεστικό οργανισμό αυτών των ε, διαδρόμων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω και εγώ με όσους επένδυσαν την ε, Επιτροπή για ένα κείμενο το οποίο αποτελεί καλή βάση για τις ε, συζητήσεις μας εδώ πέρα και ακούγοντας τώρα βεβαίως και αυτά τα οποία είχε πει το Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε το τι γίνεται, παραδείγματο χάρη, με την χρηματοδότηση ασφαλών ε, θέσεων στάθμευσης ε, κατά μήκο των αυτοκινητοδρόμων, ε, κάτι το οποίο τώρα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Επίση, θα πρέπει να δούμε και το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, όπου δεν βλέπω μια ολοκληρωμένη σκέψη για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι τέτοιο. Θα πρέπει νομίζω να ε, υπάρξει μια θέση για αυτό το ε, κομμάτι και στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε την ε, δια σύνδεση των λιμανιών που είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι επίσης υποχρεωτικό όταν μιλάμε για την εσωτερική ναυσιπλοεία να υπάρχει υποχρέωση και υπάρχει υποχρέωση των λιμανιών να συνδέονται με τους σιδηροδρόμους, αλλά όχι αντιστρόφως. Οι σιδηρόδρομοι δεν υποχρεώνονται να πηγαίνουν μέχρι τα λιμάνια. Και όταν μιλάμε για εσωτερικούς ε, λιμένες, δεν είναι σαφές το ποιοι λιμένες εντάσσονται στο συνελικό ε, δίκτυο και το εάν αποτελούν καν εσωτερικοί λιμένες ε, μέρος του δικτύου του βασικού. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί αν δούμε το σημερινό προϋπολογισμό των διευρωπαϊκών δικτύων μέχρι το 2013, μιλάμε για ποσοστό μικρότερο του 1% ε, ενώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό εκεί πέρα. Αυτά και οπωσδήποτε θα τα ξαναπώ και στην περαιτέρω συζήτηση. Ε, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Συμφωνώ με τη δημιουργία του κεντρικού, του βασικού δικτύου και του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και συμφωνώ με τις διασυνοριακές διασυνδέσεις που προτείνονται. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να καθορίσουμε με καλύτερο τρόπο τους βασικούς στόχους και τα βασικά κριτήρια. Σε σχέση με τον κανονισμό διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής, βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί και τα οποία θέτουν τοπικές και περιφερειακές αρχές. Δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε τα ερωτήματα αυτά. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να τους δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Τώρα, όσον αφορά τη μεθοδολογία, θα πρέπει να συζητήσουμε σε ποιο βαθμό η μεθοδολογία αντανακλά τελικά τα διασυνοριακά και κοινωνιολογικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και γειτονικών κρατών. Επίσης πρέπει να δούμε πώς θα καλυφθεί η Τσεχία και πώς θα διασυνδεθεί όχι μόνο με τη Γερμανία αλλά και με τη Σλοβακία. Και θα πρέπει επίσης να καταφέρουμε να δούμε πώς θα ορίσουμε αυτό το οποίο αποκαλούμε μεγάλες πόλεις. Επίσης, ποια είναι η προστιθέμενη αξία όλου αυτού του εγχειρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να καθοριστεί καλύτερα, γιατί συνδέεται με τον ορισμό που χρησιμοποιούμε για ένα έργο, για ένα σχέδιο κοινού συμφέροντος. Να αναφερθώ σε κάποια έργα τα οποία λαμβάνουν χώρα, προετοιμάζονται στα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ συχνά δεν έχουμε την απαραίτητη εμπειρία κατά την προετοιμασία των έργων αυτών. Και υπάρχουν λοιπόν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία αναγκάζονται να προσφύγουν σε πολύ ακριβές εταιρείες παροχής τεχνικών συμβουλών. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με ένα τέτοιο κόστος. Τώρα, η αρχή use it or lose it, απώλεια σε περίπτωση μη χρήσης θα μπορούσαν κάποια κράτη-μέλη να ενθαρρυνθούν να συμμορφωθούν με την αρχή αυτή, προκειμένου εξ αρχής να υποβάλουν κάποια ποιοτικά σχέδια τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ή από κάποιο άλλο μέσο. Όσον αφορά τώρα τα διασυνοριακά έργα, ο ρόλος των συντονιστών θα πρέπει να ενισχυθεί και ρόλος τους θα πρέπει να είναι να μειωθεί το διοικητικό άκθος και να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι θα πρέπει μέσω νέας μεθοδολογίας τεντή να δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε τις υποδομές μεταξύ κρατών μελών και ένα πλαίσιο διασύνδεσιμότητας και να διασφαλίσουμε διατροπικές διασύνδεσεις να ορίσουμε την εσωτερική ναυσιπλοεία μέσα στα πλαίσια του ΤΕΝΤΗ και τη συνδεσιμότητα λιμένων. Θα ήθελα να σας πω ότι η Ανατολική Ευρώπη και στα νέα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουμε και τις οδικές υποδομές, διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, ποιοτική διαφορά μεταξύ κρατών μελών ως προς, την, ε, ως προς τις μεταφορές θα πρέπει να δούμε πώς ορίζουμε τις ε, μεθοδολογίες μας, γιατί για λόγους διαφάνειας θα πρέπει η μεθοδολογία να συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό. Επίσης το παράρτημα 3 μας δίνει την χαρτογράφηση ε, σε σχέση με τις γειτονικέ χώρες. Και νομίζω ότι ένα κομβικό σημείο είναι πολύ λίγο για μία χώρα, γιατί εμείς έχουμε ε, συνορεύουμε με την Ουκρανία και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη διαφορετικούς ε, τύπους μεταφορών. μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, μεγάλης ακτίνας συνόρων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όταν μιλάμε για ένα επεκτεταμένο δίκτυο μέχρι το 2020 ή 2030 θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι περιφέρειες σε αυτή την ε, ε χαρτογράφηση στο ε, Γαλάτιο, Μπραήλα και Ματσίν υπάρχουν, υπάρχει διατροπική, υπάρχουν διατροφ, διατροπικές μεταφορές και μέσω Δούναβη με την Μαύρη Θάλασσα και μέσω σιδηροδρομικών μεταφορών. Πρόεδρος, θα ήθελα να πω κι εγώ μερικά πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σκόπιμο να πω ότι θα ενθαρρύνω τους δύο συνεισηγητές γιατί μιλήσαμε για τα ΤΕΝ και για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αλλά βλέπω ότι έχουμε και μία ε, προσέγγιση shopping list γιατί όταν προβήκαμε στα πρώτα τεν εγώ ήμουνα εδώ και τι έκανε η Επιτροπή χαρτογραφήσεις και μόνο και τίποτα άλλο. Και όταν κανείς παρουσιάσει ένα χάρτη σε ένα κράτος μέλος, τι κάνει. Απλώς τραβάει γραμμές ε, δόθεν κακήθεν για σημεία σύνδεσης. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στα ε, κράτη-μέλη ότι μιλάμε για TEN-T. Υπάρχει και ένα E ενδιάμεσο που σημαίνει European. Δεν μιλάμε για εθνικά ε, δίκτυα, μιλάμε για ευρωπαϊκά δίκτυα. Άρα η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να είναι η μείζων προτεραιότητά μας. Αν θέλουν τα κράτη-μέλη να κάνουν ε, οδικές ε, αρτηρίες ε, ή σιδηροδρομικές μεταφορές ή εσωτερικές, εσωτερική ναυσιπλοεία, ας το κάνουν για τη χώρα τους αλλά ε, αν μιλάμε για διευρωπαϊκά δίκτυα, τότε φέρουν και ένα βάρος, ένα ειδικό βάρος, για να ορίσουν προτεραιότητες ευρωπαϊκού επίπεδου και όχι μόνο εθνικού. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα δοθεί μάχη όχι εδώ μεταξύ ημών, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι κινούμαστε προς ε, τη σωστή κατεύθυνση. Ας βγάλουμε τη μαύρη τρύπα της τσεχικής δημοκρατίας, όπως είπε ο Γιάννα, και δεν συμφωνώ μαζί του. Έχουμε τις παραμέτρους για το πού πάμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Όμως θα δοθεί μεγάλη μάχη σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών. Ας μην έχουμε καμία αυταπάτη περί αυτού. και οι δύο οι συγητές έχουν ένα δύσκολο ε, έργο στα τέντη. Τι θα κάνουν οι κύριοι Ρίκε και Γιάλα Σέντερ όταν αρχίσουμε να μιλάμε για χρήματα. Για... Γιατί μπορώ να σας πω ότι ως προς τα ταμεία, το Ταμείο Συνοχής μου λένε ήδη ότι τους αποσύρουμε τα χρήματα. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη. Να δούμε δηλαδή τι θέλουμε εμείς για τα ten Ελπίζω οι εισηγητές και με, το, ε, και με το μέσο Connecting Europe και με το ten να είναι ε, αρκετά υπομονετικοί έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα συνεπές έργο. Να υποστηρίξουμε λοιπόν τους εισηγητές έτσι ώστε να έχουμε συνεκτική θέση του Κοινοβουλίου. Ωραία. Ο κύριος Πακέ έχει το λόγο. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και κάποιος άλλος, κύριε Πακέ. Και στο τέλος οι δύο συνεισηγητές. Λοιπόν, η Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά πράγματα υπόθηκαν από τους ίδιους τους Ευρωβουλευτές. Δύο ερωτήματα θέσατε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας απαντήσουμε και γραπτός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και χαίρομαι πάρα πολύ για την εργασία που έχει γίνει από τους συνσηγητές, από τους σκιώδεις και από τα υπόλοιπα μέλη. Βλέπετε ποια είναι η βασική πρόκληση, την κατονείται πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική υποδομών που αποτελεί πραγματικά την ραχοκοκαλιά της εσωτερικής αγοράς. Θέλουμε να έχουμε ένα πολυτροπικό μοντέλο για την εσωτερική αγορά αλλά αυτή η βασική υποδομή που θα δημιουργήσει τον διευρωπαϊκό χώρο μεταφορών απαιτεί ουσιαστικά τη δέσμευση των κρατών μελών, αλλά και τη δέσμευση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες, ξεκινώντας από την υφιστάμενη υποδομή, την οποία θα πρέπει να βελτιώσουμε. Αυτό είναι το βασικό πνεύμα της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή σας και γενικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει με την πρόταση αυτή κατά τη διάρκεια της συναπόφασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να συμβάλλει στην ακρόαση την οποία θέλουν να διοργανώσουν οι συνεισηγητές τον Μάιο Νομίζω ότι τα τρία ζητήματα, μεθοδολογία, το κεντρικό δίκτυο των διαδρόμων, καθώς επίσης και οι απαιτήσει για το κεντρικό δίκτυο και το εκταμένο δίκτυο, τα τρία αυτά ζητήματα αποτελούν και τα κεντρικά σημεία της ε, πρότασης. Ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω και αν χρειάζεστε περισσότερε εξηγήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε στη διάθεσή σα. Προσβλέπουμε λοιπόν σε μια θετική συνεργασία με του συνσηγητέ του επόμενου αυτού μήνε οι οποίοι όντως θα είναι δύσκολοι όχι στη συζήτηση που θα κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά στη συζήτηση που θα πρέπει να κάνουμε και συνεργασία που θα έχουμε με το Συμβούλιο. Δεν είναι πολύ εύκολο να καταφέρουμε να περάσουμε και στα υπόλοιπα α, θεσμικά όργανα τη συμφωνία που έχουμε εδώ πέρα. Γιώργο, θέλει εσύ να ξεκινήσει τώρα πρώτος και συνέχεια θα μιλήσει και ο Ισμαήλ. Ε, thank you, Chair. Um... Θα ήθελα να τους συναδέλφους, τους σκιώδεις συζητητέ και τους άλλους συναδέλφους που πήραν ε, το λόγο. Ακούστηκαν ε, πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να λάβουμε και εμείς υπόψη μας στη συνέχεια της εργασίας μας. Αν, αν και επιμένω στο ότι η συνεργασία αυτή θα είναι συνεχής και ουσιαστική και αυτή είναι μια δέσμευσή μας και εμού και του ε, κυρίου Ερτούγκ. Όσον αφορά ορισμένα ερωτήματα που ετέθησαν απευθείας ε, σε μένα, ε, θα ήθελα να δώσω πολύ γρήγορα κάποιες απαντήσεις, αν και ειδικά με την κυρία Γιάλα Σέντερ θα έχουμε πολλές ευκαιρίες στην επικοινωνία που θα έχουμε, γιατί και εκείνη είναι συνεισηγητής στο Connecting Europe Facility, επομένως όπως είπα και στην αρχή, οι συναντήσεις οι δικές μας με τους ε, δύο συνεισηγητές του Connecting Europe Facility θα είναι συνεχής. Και επομένως θα έχουμε πολλές ευκαιρίες είτε στο πλαίσιο της Επιτροπής είτε κατηδία να τα συζητήσουμε. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα, κυρίως με ρώτησε για, τις, ε, για τα deadlines, για τα χρονικά όρια, κατά πόσο υπάρχει ευελιξία ή όχι και τι σημαίνει ευελιξία για μένα προσωπικά δεν υπάρχει πρόβλημα και νομίζω και για τον ε, Ισμαήλ δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να δεχθούμε το 2030 και το 2050 ως ε, όρια. Και εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ζητούν ε, μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τα χρονοδιαγράμματα. Εκεί νομίζω ότι το βασικό αντεπιχείρημα σε όσοι ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία είναι ότι ίδια, ε, ήδη το σχέδιο του κανονισμού προβλέπει μία αναθεώρηση το 2023. Επομένως, εάν τα πράγματα μέχρι το 2023, εάν έχουμε ε, εντοπιστεί είτε δυσκολίες, είτε αδυναμίες υλοποίησης, είτε άλλα προβλήματα, υπάρχει το 2023 για να τα ξαναδούμε. Επομένως, θέση μου είναι ότι το 2003 το 2030 και το 2050 είναι επαρκή χρονικά όρια για να προχωρήσουμε. Αλλά η ευελιξία, η προβλεπόμενη ευελιξία, και αυτή θα ήταν η απάντησή μου στη βασικό της ερώτημα, είναι ότι το 2023 προβλέπεται μια, έτσι κι αλλιώς, μια ε, αναθεώρηση. Για το use it or lose it. Ε, θεωρώ ότι εάν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε επιτέλους με την εφαρμογή αυτού του μεγάλου σχεδίου, για την ενοποίηση των μεταφορών στην Ευρώπη. Ουσιαστικά την, ε, την το σύστημα αιμοδοσίας της ενίας αγοράς. Εάν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε, πρέπει να είμαστε αρκετά αυστηροί με την εφαρμογή και την αξιοποίηση της χρηματοδότησης. Ε, βεβαίως, η διατύπωση από μόνη της είναι πάρα πολύ αυστηρή. Χρησιμοποίησέ τα ή τα χάνεις. Ενδεχομένως εδώ θα πρέπει να δούμε κατά πόσον τα χρήματα αυτά θα επιστρέφουν στην δεξαμενή των χρημάτων ε, που προβλέπονται για χρηματοδοτήσεις και αν το κράτος που τα έχει χάσει σε πρώτη φάση έχει τη δυνατότητα, αφού κάνει κάποιες διορθώσεις και αφού δώσει κάποιες εγγύησεις, να τα ξαναδιεκδικήσει στο μέλλον. Αυτό θα ήταν μια πιθανή διέξοδος που θα έκανε αυτή την αρχή λιγάκι πιο ρεαλιστική και πιο ευέλικτη. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία θα δούμε στην πορεία των συζητήσεών μας. Ε, τώρα όσον αφορά για τους, ε, για τους διαδρόμους, ε, πράγματι πιστεύω ότι οι διάδρομοι από τη φύση τους ε, θα, είναι, θα πρέπει να ήταν κυρίως ενταγμένοι στο guidelines, στον ε, κανονισμό για τις κατευθυντήριες γραμμές και λιγότερο στο Connecting Europe Facility. Αλλά αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δούμε, αλλά μεθοδολογικά, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανάλυση του τι είναι διάδρομος πώς εφαρμόζεται, ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο των guidelines. Αλλά εγώ δεν θέλω τώρα να εισάγω ένα σημείο τριβής μεταξύ των εισηγητών των κατευθυντηρίων αρχών και του Connecting Euro Facility, αλλά είναι μια σκέψη που νομίζω ότι έχει αρκετή βάση, την οποία πάντως ε, μπορούμε να δούμε. Ε, αυτές σε αυτό το στάδιο θα μπορούσαν να είναι κάποιες γενικές απαντήσεις. Συγκράτησα με ενδιαφέρον την περίπτωση της Λιέγης, αλλά όλα αυτά όπως σας είπα είναι η πρώτη συζήτηση. Θα έχουμε πολύ χρόνο, πολλές συναντήσεις, πολλές και ε, εξαντλητικές ανταλλαγές απόψεων ε, στον επόμενο, στον επόμενο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Κουμουτσάκο. Κύριε Σερτού, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους και εγώ για τις παρεμβάσεις τους να τονίσω ακόμη μια φορά πως είναι αποφασιστική σημασία εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε μια ισχυρή θέση έναντι του Συμβουλίου και θέλω να επαναλάβω πως εμείς στο Κοινοβούλιο θα, θα βρούμε μια λύση, αυτό θα γίνει. Αλλά παρόλα αυτά τα επίμαχα σημεία είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν με το Συμβούλιο και όχι με τους συναδέλφους εδώ στο Κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά να υπενθυμίσω γιατί δεν αναφέρθηκε. Πώς προέκυψε η πρόταση της Κομισιόν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και να το λέμε αυτό και στις εθνικές συζητήσεις πως ε, υπήρξε μία φάση δύο ετών όπου τα κράτη-μέλη σε διάφορες επιτροπές είχαν δυνατότητα να συνεισφέρουν στη δημόσια διαβούλευση. Και από εκεί προέκυψε ο πυρήνας και αυτό θα πρέπει να το πούμε και στο Συμβούλιο Υπουργών. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να τονίσω τρία ε, σημεία ε, για αυτά τα οποία είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ για τις πράξεις ε, κατεξιοδότηση ανέφερα πως θα πρέπει να συζητήσουμε το εάν και πως θα είναι δυνατόν να μπορούμε να διαλέγουμε έργα τα οποία θα ανταποκρίνονται και στη μεθοδολογία μας. Και εάν ναι, πώς θα πρέπει να γίνουν. Και βεβαίω σημαντικό είναι όταν μιλάμε για τις πράξεις κατεξιοδότηση, τουλάχιστον να συμφωνήσουμε στο ότι δεν μπορεί να είναι δυνατόν να υπάρξει κάποια αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το Κοινοβούλιο. Αλλά νομίζω πως αυτό αφορά πολύ περισσότερο νομοθετική διαδικασία παρά τις πράξεις αυτές. Τώρα για την εκτελεστική αυτή υπηρεσία που ανέφερε η κυρία Γιάλα Σέντερ και αυτό είναι σημαντικό και σχετίζεται με τους διαδρόμους και τις πλατφόρμες ε, των διαδρόμων και εκεί πέρα πρέπει να συζητήσουμε. Εγώ δεν θα ήμουν κατά του να δοθούν περισσότερε αρμοδιότητε στην εκτελεστική αυτή υπηρεσία για να επιτύχουμε το στόχο αυτό γρηγορότερα. Αλλά να αναφερθώ ακόμη μια φορά στην διαφάνεια και στην υποχρέωση πληροφόρηση της Κομισιόν, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για το δικό του ε, συμφέρον. Και δεν ξέρω, δεν είναι σωστό νομίζω να περιμένουμε μέχρι τον ε, Μάιο και την ακρόαση για να ακούσουμε πληροφορίες. Θα περάσουν τρεις μήνες μέχρι τότε. Θα σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα και πιθανώς ε, να προκύψουν και κάποιες ε, νέες ιδέες που δεν ξέρουμε κατά πόσον θα είναι παραγωγικές. Θεωρώ λοιπόν πως πριν την ακρόαση θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει η μεθοδολογία και τι εννοούμε με αυτήν. Κάτι άλλο επίσης ε, σημαντικό που αναφέρεται και στο Συμβούλιο αλλά και στους ε, συναδέλφους που ε, ανησυχούν ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση των ταμείων συνοχής και η χρηματοδότηση θα πρέπει να τονιστεί γιατί δεν είναι κατά την άποψή μου ξεκάθαρα το τι εννοούμε με αυτή την αρχή το, το use it or lose it. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή, θα χάσουν τα κράτη-μέλη τα λεφτά. Αν, αν τα χάσουν τι γίνεται μετά, τι πρέπει να κάνουν για να μην τα χάσουν. Όλα αυτά είναι θέματα που ενδιαφέρουν τους ε, συναδέλφους και θα αποτελέσουν βεβαίω και το κριτήριο για την αποδοχή από τα εθνικά κοινοβούλια και κάτι ακόμα διάδρομοι και πλατφόρμες να το ξαναπώ πολλά πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι ρόλο θα παίζει ακριβώς θα παίζουν οι συντονιστές κάποια σαφήνεια υπάρχει στα άρθρα, αλλά νομίζω θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το ζήτημα και οπωσδήποτε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και διαφάνεια. Κατά λοιπά, είμαι ικανοποιημένος και ευχαριστώ ε, τους συναδέλφους για την κριτική ματιά ε, με την οποία είδαν αυτό το θέμα και οπωσδήποτε θα το δουν και τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και για την πειθαρχία τους, για το ότι δεν ξεπεράσαμε το χρόνο τηρήσαμε το χρονοδιάγραμμα. Επαναλαμβάνω πως πρόκειται για την αρχή ε, μιας διαδικασίας. Θα έχουμε έξι μήνες ε, μπροστά μας μέχρι να φτάσουμε, τουλάχιστον έξι μήνες μέχρι να φτάσουμε στην ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Οπότε σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση και να σας υπενθυμίσω πως αύριο το πρωί στις 9 ε, θα ψηφίσουμε την έκθεση Taylor, οπότε φέρτε τις κάρτες σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και